Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Ενώ συνεδριάζουν κάποιοι ακόμα με την Επιτροπή Εσωτερικών, εμείς καλωσορίζουμε εδώ τους συναδέλφους από την Επιτροπή Εξωτερικών και την Επιτροπή Ανάπτυξης. Καλωσορίσατε για να ακούσουμε την ειδική έκθεση για την Τουρκία από ε, την, ε, το ελεκτικό συνέδριο. Ε, κύριε Μακάλιστερ, θέλετε να πείτε δύο λόγια εισαγωγικά και υποδοχής. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητή κυρία Γκρέσλε. Θέλω να σας καλωσορίσω όλους στην παρουσίαση της έκθεσης, ειδικής έκθεσης για την Τουρκία. Καλό είναι που συνεδριάζουμε πέρα από όρια επιτροπών Καλωσορίζω την εργασία του ελεκτικού συνεδρίου. Το Κοινοβούλιο τη λαμβάνει σοβαρά υπόψη κατά τον κοινοβουλευτικό του έλεγχο. Σε ό,τι αφορά την πρώτη έκθεση για τη διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία, είναι πολύ επίκαιρη γιατί εμείς θα συζητήσουμε την 28η ε, έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία το Φεβρουάριο, στις 4 του μηνός το ταμείο αυτό ήταν πάρα πολύ χρήσιμο ε, γιατί ανταποκρίθηκε στην κρίση και στις πρώτες ανάγκες στις πιο οξύες των προσφύγων. Ευχαριστώ η κυρία Μακάβαν. Ευχαριστώ, Ντέιβιτ, και ευχαριστώ και εσά, κυρία Γκρέσλε, και την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού για τη σημερινή κοινή συνεδρίαση. Είναι τρει σημαντικέ εκθέσει για την δική μα Επιτροπή. Η πρώτη είναι για την Τουρκία το 2015 έχω πάει, είχα πάει στην Τουρκία, στο Gaziantep, πριν δημιουργηθεί αυτή η διευκόλυνση και είδα τι συμβαίνει ε, εκεί. Η δική μας επιτροπή σε τρεις εβδομάδες θα μεταβεί ξανά στο Gaziantep για να δει τι έχει γίνει και περιμένουμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακούσουμε ποια είναι τα διδάγματα και τι πρέπει να γίνει ακόμα. Για το καταπαστηματικό ταμείο για την Αφρική και πάλι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για ποιο λόγο γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίρνει πολλά χρήματα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη που ήταν προγραμματισμένα για διάφορα κράτη και τα πηγαίνει στην Αφρική. Και τα σπαίνει σε μια σειρά προγραμμάτων. Ε, το Κοινοβούλιο ήταν επιφυλακτικό για την ίδρυση αυτού του καταπιστευματικού ταμείου και πώς ε, δαπανώνται τα κονδύλια και η Επιτροπή Ανάπτυξης ήταν πάρα πολύ ανήσυχη και ήθελε τα χρήματα αυτά να πηγαίνουν για την ανάπτυξη. Για την ανάπτυξη επαναλαμβάνω, γιατί από εκεί τα πήραμε και δεν είναι τα λεφτά αυτά για να χτίζουμε ή για να εκτοπίζουμε και να επαναπατρίζουμε ε, αναγκαστικά ε, ανθρώπους στην Αφρική. Ξέρουμε ότι υπάρχουν νέες ανάγκες Αυτή τη στιγμή συζητούμε ένα άλλο ταμείο που μπορεί να είναι κάπως διαφορετικό από το γενικότερο κατεπαστηματικό. και εμείς ε, ε, κυβερνητικέ οργανώσεις ε, δίνουν ε, βοήθεια ανθρωπιστική, είναι πάρα πολύ χρήσιμοι συνομιλητέ, και πραγματικά θέλω πολύ και με ενδιαφέρει να ακούσω τι έχετε να πείτε για την ανθρωπιστική αυτή χρήση και την αναπτυξιακή βοήθεια προς τη ΜΚΙΟ. Ευχαριστώ. Θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Γιάκοψεν για να μας παρουσιάσει την έκθεση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε, κύριε Συμπρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να σας παρουσιάσω την ειδική έκθεση για τη διευκολύνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία. Θα σας παρουσιάσω τα κύρια ευρήματα, τα συμπεράσματα και τις συστάσεις ε, όπως προκύπτουν από τον έλεγχό μας. Λόγω της θέση της, η Τουρκία είναι χώρα και υποδοχής ε, και διέλευσης για πολλούς ε, πρόσφυγες που έρχονται από περιοχές ε, συγκρούσεων στην περιοχή λόγω της πίεση των μεταναστευτικών ροών, λόγω του πολέμου στη Συρία. Έχει η Τουρκία φιλοξενούμενο το μεγαλύτερο πληθυσμό προσφύγων στον κόσμο, σχεδόν 4 εκατομμύρια, 3,5 εκατομμύρια Σύρους και από την έναρξη της κρίσης η Τουρκία παρήχε συνεχή σημαντική υποστήριξη προς τους πρόσφυγες. Η διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία έχει αρχικό προπολογισμό 3 δισεκατομμύρια ε, ευρώ που θα χρησιμοποιούνταν το 2016 και το 2017. Αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι από αυτό το ποτό είχαμε το μισό προπολογισμό από τα κράτη-μέλη και τον άλλο μισό από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Το 2018 το Συμβούλιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να στείλει τη δεύτερη δόση και πρόσθεσε επιπλέον 3 δισεκατομμύρια ευρώ χρηματοδότηση στον προπολογισμό τη διευκόλυνση προ ε, δαπάνη για το 2018 και 2019. Στόχος ε, είναι η ο συντονισμό των δράσεων που χρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό και από τι ε, συμμετοχέ των κρατών μελών και η βελτίωση τη αποτελεσματικότητα και τη συμπληρωματικότητα που ε, παρέχεται στους πρόσφυγες ε, στην Τουρκία και στου μετανάστες. Τι ζητήματα εξετάσαμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Εξετάσαμε κατά πόσο από η διευκόλυνση υποστήριξε αποτελεσματικά τους πρόσφυγες στην Τουρκία. Εστιαστήκαμε στη διαχείριση του πρώτου τμήματος της ε, διευκόλυνσης και στα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στο ανθρωπιστικό σκέλος. Πρώτα απ' όλα εξετάσαμε κατά πόσο η δομή και η λειτουργία αυτής της διευκόλυνσης ως μηχανισμού συνέβαλε σε σημαντική και καλά συντονισμένη και γρήγορη υποστήριξη. Δεύτερον, εξετάσαμε το κατά πόσο τα ανθρωπιστικά έργα τα οποία χρηματοδότησε η διευκόλυνση επέτυχαν τα αποτελέσματα που είχαν σχεδιαστεί αυτό βάσει ενός δείγματος 10 ανθρωπιστικών έργων ε, ύψους ε, άνω των 300 ε, εκατομμυρίων ευρώ. Τι βρήκαμε συνολικά το μήνυμα της έκθεσης είναι ότι υπό τις δύσκολες συνθήκες η διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία κινητοποίησε γρήγορα αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ από τα κράτη-μέλη και τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό ως μια γρήγορη απάντηση στην κρίση των προσφύγων. Ωστόσο δεν πέτυχε τους στόχους αποτελεσματικού συντονισμού αυτής της ε, απόκρισης. Το έργο που ελέγξαμε παρήχε επαρκή υποστήριξη στους ε, πρόσφυγες. Αυτό σημαίνει ότι τα περισσότερα έργα πέτυχαν τα αποτελέσματά τους. Για παράδειγμα, το έργο ε, κοινωνικής προστασίας ε, έκτακτης ανάγκης για τις καθημερινέ ανάγκες του 1,3 εκατομμυρίων προσφύγων στην Τουρκία. Από την άλλη, το μισό έργο δεν είχε επιτύχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και 9 από τα 10 έργα χρειάστηκε να παραταθούν. Όταν μιλάμε για αποτελέσματα, συνήθως αναφερόμαστε σε κάτι που μακροχρόνια να έχει υποφελεί αποτελέσματα που μπορούν να ε, λειτουργούν αυτόνομα χωρίς περαιτέρω ε, οικονομική υποστήριξη. Το δύσκολο περιβάλλον ήταν το κύριο εμπόδιο που είχαμε στη σωστή διαχείριση των έργων. Επίσης προσδιορίσαμε περιθώριο βελτίωσης τη αποτελεσματικότητα των έργων. Επί παραδείγματι, κατά την αναθεώρηση των προτάσεων για έργα, η Κομισιόν δεν έδειξε συνέχεια και αποτελεσματικότητα στην αξιολόγηση του κατά πόσο ήταν τα κόστη λογικά. Επίση, όσον αφορά τα πάνε ε, για του εταίρου ε, οι οποίοι εφαρμόσαν τα διάφορα επιμέρου έργα, θεωρήσαμε ότι ήταν υψηλό και κάποιε πληρωμέ δεν συμφωνούσαν με τι πραγματικέ εκροέ μετρητών. Όσον αφορά τα έργα υποστηρίξη σε μετρητά, όσον αφορά τη διευκολύνση κομισιών εντόψη τη ε, κατά προτεραιότητα ανάγκη των προσφύγων βάσει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση αναγκών. Ωστόσο, αυτή η συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των αναγκών σε αστικές υποδομές και κοινωνικο-οικονομική υποστήριξη είχε ως αποτέλεσμα ότι δεν καλύφθηκαν επαρκώς αυτοί οι τομείς. Η διευκόλυνση υποστήριξε παρόμοιες δραστηριότητες στους τομείς της υγείας και της παιδείας μέσω διαφόρων εργαλείων. Έτσι κατέστη ο συντονισμός πιο περίπλοκος με αποτέλεσμα την εσωτερική χρήση διαφορετικών διαχειριστικών δομών για τη χρηματοδότηση παρεμφερών έργων. Παρότι έχουμε εντοπίσει κάποια καλά παραδείγματα στον τομέα της υγείας όπου η Κομισιόν υποστήριξε την μετάβαση από την ανθρωπιστική σε πιο βιώσιμη υποστήριξη και βοήθεια, αυτή η συμπληρωματικότητα δεν ε, ε, επετεύχθη συστηματικά. Η Κομισιόν ε, εφάρμοσε μέτρα παρακολούθησης των ανθρωπιστικών έργων και βασικό εμπόδιο ήταν οι τουρκικές αρχές, οι οποίες αρνήθηκαν την πρόσβαση σε στοιχεία δικαιούχων για τα δύο έργα υποστήριξης με μετρητά. Και στην πραγματικότητα ούτε η Κομισιόν ούτε εμείς ως ελεγκτές καταφέραμε να βρούμε τους δικαιούχους των έργων από την εγγραφή τους μέχρι την πληρωμή. Και αν ελεγκτή αυτή η κατάσταση αποτελεί σοβαρό πρόβλημα όταν δεν μπορεί να παρακολουθεί την πορεία μιας πληρωμής το πλαίσιο πόρων της διευκολύνσης ε, ε, δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμα για να αναφερθούν οι πόροι. Αυτό σημαίνει ότι τα σημεία αναφορά, ποσοτικοποιημένοι στόχοι κτλ. δεν είχαν ολοκληρωθεί όταν κάναμε τον έλεγχο. Ανακαλύψαμε ότι οι δημόσιε εκθέσει ήταν περιορισμένε και το αντικείμενό του δεν κάλυπτε ολόκληρη την υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ του πρόσφυγε στην Τουρκία. Ο συμπέρασμα λοιπόν, η διευκόλυνση βοήθησε σημαντικά, αλλά απαιτούνται βελτιώσει για καλύτερη, ψηλότερη αξία για τα χρήματα που έχουν δοθεί. Τι συνιστάμε εμεί ω ελεγκτέ. Η έκθεσή μα περιλαμβάνει διάφορες συστάσει που πιστεύουμε θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη βελτίωση τη αποτελεσματικότητα κατά την υλοποίηση του δεύτερου κομματιού του προπολογισμού τη διευκόλυνση, Προτείνουμε λοιπόν να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι ανάγκε των μεταναστών για την κοινωνικο-οικονομική του υποστήριξη να βελτιωθεί η απλούστευση και η συμπληρωματικότητα της υποστήριξης, να υλοποιηθεί μια στρατηγική για τη μετάβαση από ανθρωπιστική σε αναπτυξιακή βοήθεια, βελτίωση της αποτελεσματικότητας των έργων υποστήριξης σε μετρητά, συζήτηση με τις τουρκικές αρχές για τη βελτίωση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος για τη ΜΚΟ και τέλος περισσότερη παρακολούθηση και, και εκθέσεις για την βοήθεια που παρέχεται στους πρόσφυγες στην Τουρκία. Η Κομισιόν δέχτηκε όλες μας τις συστάσεις και θέλω να του ευχαριστήσω για την επικοδομική του βοήθεια και συνεργασία κατά τους ελέγχους. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ να απαντήσω σε οποιασδήποτε ερωτήσεις έχετε για την έκθεση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Η συγγετριά μα που είναι η κυρία Κινίτση, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε να χαιρετήσω τους συναδέλφους ε, της ΑΦΕΤ και της ΔΕΒΕ, να ευχαριστήσω την κυρία Γιάκοψεν και το Ενεκτικό Συνέδριο για την ειδική έκθεση για την διευκόλυνση για τους πρόσφυγες ε, στην Τουρκία. Το μέσον αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά της, του κοινού σχεδίου δράσεως ε, της, 10, της 5 Οκτωβρίου 2015 μεταξύ των κρατών μελών και της Τουρκίας στο πλαίσιο δηλαδή, της συμφωνίας του 2016. Το μέσο ήταν κάπως αντιφατικό υπό κάποια σημεία νομικής και πολιτικής εξέτασης, αλλά κινητοποιεί και συντονίζει τις, ε, τους χρηματοδοτικούς πόρους του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κράτων μελών για τους άνω των 4 εκατομμύρια πρόσφυγες που φιλοξενεί η Τουρκία στο εδαφός της από την Ιρακινή κρίση και μετά. Τώρα, σχετικά με τις απορίες, ε, σχετικά με το statement, μιλούμε εδώ για μια ανθρωπιστική στόχευση, ε, την οποία μπορεί να υποστηρίξει κανείς και επί της οποίας ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να διατηρούν υψηλή την προσοχή τους για να είναι αποτελεσματικό το μέσο έτσι όπως σχεδιάστηκε. Ή στην πλαίσιο του ελέγχου του προϋπολογισμού Ακούσαμε το ποσό, τα αρχικά 3 δισεκατομμύρια και μια δεύτερη δέσμη 3 ακόμα δισεκατομμύριων τον περασμένο Ιούνιο. Όλα αυτά ε, απαιτούν μια ιδιαίτερη προσοχή και μια ιδιαίτερη παρακολούθηση. Και η ιστορική αυτή θα πρέπει να σημειώσουμε θετικά, όπως μόλις σημειώσαμε και το ελεγκτικό συνέδριο, ότι το μέσον έχει καλύψει στις βασικές του ανάγκες τα κενά και την υποστήριξη που έπρεπε να δώσουμε στους πρόσφυγες. Τώρα, για τις ε, συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου, ε, εστιαστήκαμε περισσότερο στην παρακολούθηση των έργων και την αξιολόγηση των αναγκών. Και επ' αυτού θα ήθελα να πω δύο λόγια. Αναφέρομαι τώρα στην απαγόρευση των τουρκικών αρχών για την πρόσβαση στον στα δεδομένα των δικαιούχων για βοήθεια και αυτό ακόμα και έναντι του ελεγκτικού συνεδρίου, επί τη βάση δηλαδή του ελέγχου που διενήργησε, σχετικά με την προστασία των ενδομένων υπό την τουρκική νομοθεσία. Τώρα, δεδομένης της ε, σημασίας των, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των προσφύγων, δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν τέτοιες δεσμεύσεις, τέτοια εμπόδια προς την ελεκτική αρχή και επομένως αυτό το θέμα θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε μαζί με τις τουρκικές αρχές ή στο πλαίσιο της υλοποίησης ακριβώς της δεύτερης καταβολής, της δεύτερης δέσμης καταβολής για το μέσον. Και θα ρωτούσα ποια βήματα θα μπορούσε να αναλάβει κανείς και την Επιτροπή που είναι παρούσα προς την κατεύθυνση αυτή. Κάτι ακόμα από το οποίο ελέγχθη και το οποίο εγείρει κάποιες ε, ανησυχίες. Είναι η αξιολόγηση των αναγκών, η οποία αξιολόγηση θεωρήθηκε ελλειπής από το ελεγκτικό συνέδριο και όχι επαρκώς αυστηρή σχετικά με τα δημογραφικά δεδομένα των ευάλωτων ομάδων. Αναφέρομαι ιδιαίτερα στις ε, γυναίκες, στις ε, γυναίκες χωρίς συνοδεία, στους ανηλίκους χωρίς συνοδεία. Νομίζω ότι η επικαιροποίηση και η χαρτογράφηση αυτών των δεδομένων των ευάλωτων αυτών ομάδων είναι κάτι το απολύτως απαραίτητο προκειμένου να, είναι, να έχει την νομιμοποίηση και την αποτελεσματικότητα πρέπει το μέσο αυτό. Και ρωτώ την Επιτροπή ποιε πρωτοβουλίε ελήφθησαν με τι τουρκικέ αρχέ ώστε να έχουμε αυτή την επικαιροποίηση του ευαίσθητου των ομάδων αυτών, του ευάλωτου. Υπάρχει και η αξιολόγηση μέσω του συστήματο των ΗΠΑ και παρότι το μέγιστο 7% ποσοστό ευθυγραμμίζεται με το χρηματοδοτικό πλαίσιο ε, που έχει συμφωνηθεί μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Εθνών, όπως λέει και το ελεκτικό συνέδριο, ε, η εφαρμογή αυτού του ποσοστού σε μεγάλη κλίμακα σε αυτό το δίκτυο κοινωνικής προστασίας θα μπορούσε να μην είναι απολύτως αναλογικό. Και εδώ θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή κατά πόσον έχει ξεκινήσει μια επαφή με τους εταίρους ώστε να δούμε τα έμεσα κόστη. Και συμπερασματικά θα ήθελα σύντομα να αναφερθώ στο ρόλο των ΜΚΟ. Η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου σημειώνει ένα δύσκολο περιβάλλον εργασίας για τις μη στην Τουρκία, με αρνητικό αντίκτυπο επί της υλοποίησης των έργων από πλευράς αυτών των οργανώσεων, Δεδομένης λοιπόν της περιπλοκότητας της θεσμικής ε, και της, θεσμικής, της πολιτικής μετά τις εξελίξεις του 2016 στην Τουρκία, ίσως θα έπρεπε η Επιτροπή να προαγάγει έναν υψηλού επίπεδο διάλογο με τις τουρκικές αρχές, ώστε να βελτιώσει αυτό το περιβάλλον εργασίας των ΜΚΟ, που παραμένουν πολύ σημαντικοί αεταίροι, ώστε να επιτύχουμε τις στοχεύσεις του μέσου, της διευκόλυνσης και για να παραέχουμε ε, την καλύτερη δυνατή βοήθεια στους πρόσφυγες. Αυτά συνοπτικά επί της δουλειά που έγινε. Να ευχαριστήσω όλους τους συνάδελφους για την προσοχή τους, να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο για τη δουλειά που έκανε και για τις συστάσεις προς τις οποίες συμφωνούμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, κυρία παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για αυτές τις ε, πολύτιμες εκθέσεις. Ευχαριστούμε και την Επιτροπή που όπως ξέρουμε την τελευταία διετία κατάφερε το κατόρθωτο μετά από τη σύναψη της συμφωνίας με την Τουρκία από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνησεών μας ώστε να βεβαιωθούμε ότι τα χρήματα που δίνονταν ε, θα έφερναν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Έχω πολλές ερωτήσεις. Πρώτον, όπως υπόθηκε ήδη στην παρουσίαση, δεν υπάρχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων των δικαιούχων που έλαβαν μετρητά από τα σχετικά προγράμματα. Αυτό που δεν καταλαβαίνω, από τα 3 δισεκατομμύρια που χρησιμοποίησε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό ήταν το εμβληματικό έργο, ήταν το έργο για το οποίο πάντα έκανα να παρουσιάσεις ο Επίτροπος, η Επιτροπή. Αυτό το έργο ήταν το πρώτο, το πρωταρχικό, που προβαλόταν ως το καλύτερο παράδειγμα. Στην αρχή της ε, υλοποίησης ε, ήταν γνωστό, αν ήταν γνωστό ότι δεν θα γνωρίζαμε πού θα πήγαιναν τα χρήματα, αν θα φτάνανε στους δικαιούγους, γιατί προχωρήσαμε αφού μια από τις βασικές προϋποθέσεις σύμφωνα με αυτή την έκθεση ε, ελέγχου ε, α, μια από τις βασικές προϋποθέσεις δεν ε, πληρούταν. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο συνεχίσαμε αφού ξέρουμε ότι δεν θα μπορούμε να παρακολουθούμε που πήγε το χρήμα. Η δεύτερη ερώτηση αναφέρεται και στην παράγραφο 38 για τις διοικητικές δαπάνες. Ένα μεγάλο τμήμα των χρημάτων λοιπόν χρησιμοποιείται από οργανισμού ε, των ΗΠΑ που λαμβάνουν διαχειριστικά κόστη 7% και έχουν ακουστεί διάφορε επικρίσει ε, και τις βρίσκουμε και εδώ σε αυτή την έκθεση. Και μετά, όταν μιλάμε για την Τουρκία ή κάποιον άλλο ε, εταίρο που ασχολείται με την υλοποίηση, μιλάμε για άλλο ένα 7% του κόστους. Και θέλω να ρωτήσω τους ελεγκτές, αυτό περιλαμβάνει και τα γενικά κόστη και τις γενικές δαπάνες. Ε, γιατί, συγγνώμη, εγώ δεν είμαι μέλος της Επιτροπής ε, Προπολογισμών. δεν διαβάζω την έκθεση αυτή γνωρίζοντα ε, όλες τις λεπτομέρειες. Υπάρχει και γενικά κόστη επιπλέον αυτού του 7%, αυτών των δύο 7% διότι αν ναι, μιλάμε για πολλά εκατομμύρια διοικητικό κόστος που σύμφωνα με αυτή την έκθεση ελέγχου δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται για το έργο. Τώρα, τα αναφέρθηκαν και αυτά τα τέλη ε, μεταφοράς μετρητών. Αν κατάλαβα καλά τη στιγμή που η, που, η στιγμή που στέλνει χρήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση σε έναν οργανισμό των ΟΕΕ και τη στιγμή που ο οργανισμός των ΗΠΑ τα στέλνει σε κάποιον εταίρο υλοποίησης παίρνει το 1% ως τέλος μεταφοράς ε, ο Οργανισμός των ΗΠΑ. Κατάλαβα καλά την έκθεση. Και η τρίτη ερώτηση είναι σε ένα από τα συμπεράσματά σας λέτε ότι χρειάζεται επανεκτίμηση της ανάγκης του να διατηρήσουμε τη διαχείριση της μετανάστευσης ως μια προτεραιότητα της διευκόλυνσης και διάβασα στην εκθέση ότι δύο είναι τα έργα που υλοποιήθηκαν υπό την επικεφαλίδα διαχείριση μετανάστευσης. Μιλάμε για 230 εκατομμύρια ε, ταμεία ΑΕΠΑ που αφορούσαν και συζητήσεις που έχουμε κάνει και στο παρελθόν για χρήματα ΑΕΠΑ, για την διαχείριση της μετανάστευσης, για κάποια σχετικά οχήματα κτλ. Θα μπορούσατε να μου πείτε τι είναι αυτά τα έργα και συμφωνεί η Κομισιόν ότι μήπω θα ήταν καλύτερα να μην συμπεριληφθούν σε αυτή τη διευκόνιση στο μέλλον. Ευχαριστώ. Πινκ πόνκ το κάναμε τώρα ανάμεσα στι διάφορε επιτροπέ, ο κύριο Δεχόφσκι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ως κύριο συζητητής, εγώ θα επικεντρωθώ μόνο σε κάποια πράγματα που κατά την άποψή μου χρειάζονται κάποια σχόλια και δεν ακούσαμε μέχρι τώρα. Θέλω να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο ε, και την κυρία Γιάκοψεν γιατί ήταν πάρα πολύ περιστατωμένη και αναλυτική η έκθεσή της. Τη διάβασα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έμαθα και πράγματα που δεν ήξερα πριν. Σας ευχαριστώ και για τα σχόλιά σας εκτός των άλλων. Γιατί βλέπω ότι μεταξύ των ευρωβουλευτών υπάρχουν πολλοί που εδώ και καιρό εστιάζουν στη μετανάστευση. Την ανάλυση σας τη θεωρώ πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, όσο και επίκαιρη, διότι η μετανάστευση παραμένει ε, ένα θέμα πάρα πολύ φλέγον και στις ευρωεκλογέ και νομίζω ότι θα είναι από τα δύο θέματα τα οποία θα κρίνουν τις ευρωεκλογές. Γενικώ θα έλεγα ότι το Ταμείο αυτό είναι ένα πάρα πολύ θετικό μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας για να βοηθούμε πρόσφυγες. Ακόμα και αν το δικαστήριο έχει εντοπίσει κάποιες αδυναμίες που καθιστούν αναποτελεσματικό ή λιγότερο αποτελεσματικό τον τρόπο με τον οποίο βοηθούμε. Όντως είναι εμβληματικέ αυτές οι πρωτοβουλίες ε, και τα έργα, ε, ας πούμε εκπαίδευση σύρων ε, γιατρών ή νοσηλευτικού προσωπικού για να έχουμε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη προς τους πρόσφυγες στην ίδια τους τη γλώσσα. Γενικά, νομίζω ότι η πολυτιμότερη βοήθεια που παρέχουμε είναι η βοήθεια στην εκπαίδευση. Εκεί υπάρχει και προστιθέμενη αξία και ένα δυναμικό για βιωσιμότητα. Εξεπλάγει λίγο διαβάζοντας την παράγραφο 44β, η οποία λέει ότι υπάρχει μια προμήθεια που παίρνουν εκείνοι οι οποίοι εφαρμόζουν τα προγράμματα μόνο και μόνο για να μεταφέρουν, να εμβάσουν κάποια χρήματα από την τράπεζα ε, στους ενδιαφερομένους δικαιούχους. Έτσι λέει, το έχουν εκεί έτοιμο. Αλλά αυτό είναι πραγματικά πεταμένα λεφτά από πλευράς ε, αποτελεσματικότητας του προϋπολογισμού. Εμείς έχουμε μια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου, έτσι δεν είναι. Για ποιο λόγο λοιπόν ε, εξακολουθούμε να ε, ανατρέχουμε σε όλες αυτές τις υπηρεσίες στο ΟΗΕ. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις δικές μας υπηρεσίες και τους οργανισμούς για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Όχι μόνο για το άσυλο και γενικότερα. Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού το λέει αυτό παγίωσε την τελευταία τριετία. Ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει επιτέλους για ποιο λόγο εξακολουθεί να μην χρησιμοποιεί τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες και οργανισμούς για το άσυλο. Αφού έχουμε ολόκληρο οργανισμό, γιατί δεν τον χρησιμοποιούμε, γιατί δεν τον αξιοποιούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ το ελεκτικό συνέδριο που μας έδωσε την δική του τοποθέτηση. Μια διαφημιστική ερώτηση και ίσως και προς την Κομισιόν. Υπό την οπτική του συνεδρίου επισκεφθήκατε νομίζω 10 συνολικά έργα. Κοιτώντας αν θέλετε τη χρηματοδοτική αλυσίδα σχετικά με την αποτελεσματικότητά τους. Για το αποτελεσματικό της συνεργασίας, το επιπλέον κόστος κτλ. Όμως πόσο αποτελεσματικά ήταν τα έργα αν είχατε μια τέτοια αίσθηση για στη βοήθεια που παρέχουν. Επίσης, αναφερθήκατε στο ότι 15% των κονδυλίων πηγαίνουν προς την εκπαίδευση, προς την παιδεία. Και στο, το 2015 η έλλειψη παιδείας ήταν από τα μεγαλύτερα εμπόδια και από, τις, από τα μεγαλύτερα κίνητρα να προσέλθουν στην Ευρώπη. Η έλλειψη δηλαδή παιδείας για τα παιδιά τους και εκεί είχαμε ακούσει ότι ίσως να ενσωματώνονταν στα τοπικά τουρκικά σχολεία τα παιδιά των προσφύγων. Επίσης αναφέρεστε στην χρησιμοποίηση κονδυλίων για την κατάρτιση σύρων ιατρών για την παροχή δηλαδή βοήθειας ιατροφαρμακευτικής όπως και δασκάλους ή μήπω τα παιδιά των Σύρων ε, απευθείας ενσωματώνονται σε τουρκικά σχολεία χωρί να έχει γίνει κάποια πρόβλεψη για εκπαίδευση στη γλώσσα τους. Τώρα για την μεταφορά κονδυλίων δεν είναι το παγκόσμιο επιστημιστικό πρόγραμμα που λαμβάνει αυτά τα χρήματα και όχι η τουρκική κυβέρνηση. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω με τους ενδιαμέσους πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών που δίνει κάποιες κάρτες σχετικά με τις μεταφορές των ε, μετρητών και τηρεί δεδομένα ο ΟΗΕ για τους ε, δικαιούχους, αυτούς που φέρουν αυτές τις κάρτες τέλος πάντων. Και νομίζω ότι έχει δίκιο ή κάτι. Δηλαδή ποιοι είναι τελικώς οι δικαιούχοι των καταβολών αυτών, των μεταφορών αυτών. Κυρία Λαμπάγιοβα, ευχαριστώ πρόεδρε. Η έκθεση λέγει ότι η βοήθεια που παρέχεται είναι πολύτιμη, αλλά νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια καλύτερη ε, σχέση, αν θέλετε, αξίας χρηματικής και έργου που παραδίδεται. Υπάρχει μια ε, περιπλοκότητα και δυσκολία εδώ πέρα, το οποίο έχει ενσωματώσει η Επιτροπή στην προσέγγιση της, αλλά χρειαζόμαστε να καταμετρούμε τα αποτελέσματα, τα παραδοτέα, για να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Έχω δύο ερωτήσεις. Ε, υπό την έννοια του ελέγχου του προϋπολογισμού και ίσως λίγο βαρετές, για την ενίσχυση αντιστοίχων δράσεων μέσω παραλλήλων μέσων, λέγει το ελεγκτικό συνεδρίο ότι τέτοιου είδους κατανομές καθιστούν το συντονισμό πιο περίπλοκο. Η Κομισιόν αναπαντά ότι η χρησιμοποίηση των παραλλήλων μέσων προκειμένου να επιταχυνθούν ή να επιταχυνθεί η ανταπόκριση γίνεται και αυτό το λόγο, αλλά αναρωτιέται κανείς μάλλον το διαφορικό χρόνο δεν είναι ο μοναδικός λόγος, δηλαδή χρόνο που χρειάζεται. Ποιος άλλος λόγος υπάρχει ρωτώ την Κομισιόν για την χρησιμοποίηση αυτών των παραλληλών μέσων. Για την πλήρη πρόσβαση τώρα στα δεδομένα των δικαιούχων, η Κομισιόν λέγει ότι μεταξύ των εταίρων έχει εγκαταστήσει δεδομένων των δυσκολιών το καλύτερο σύστημα που μπορούσε. Ε, ε, πώς όμως καταλήγει στο, στο συμπέρασμά της η Κομισιόν για την επιλογή τους και το συνέδριο συμφωνεί αν δηλαδή αυτά τα συστήματα ελέγχου είναι τόσο αποτελεσματικά Κάτι θα πρέπει να μας έχει διαφύγει. Συνάδελφος Αλή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Κυρία Γιάκοψεν, με όλοι ότι η διευκολύνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία αποτελεί κεντρικό στοιχείο της συμφωνίας του 2016 και ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης που ξεκίνησε το 2015 και που πλήττει την Ευρώπη. Είναι ορατή η μείωση των προσφύγων, ειδικότερα στην νότια, κεντρική και ανατολική Ευρώπη, ειδικότερα όσον αφορά τα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διευκολύνση αυτή ω μηχανισμό συντονισμού της οικονομικής ε, στήριξης Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στα γειτονικά μα κράτη-μέλη έχει δείξει γενικά καλά αποτελέσματα κατά την πρώτη φάση τα οποία αναμένουμε να συνεχιστούν με καλά αποτελέσματα και στη δεύτερη φάση. Δεν ζούμε σε ένα τέλειο κόσμο. Υπάρχουν κάποιες ελλείψεις ε, όσον αφορά την επίτευξη του συντονισμού της οικονομικής στήριξης. Γι' αυτό όμως θα ήθελα να συγχαρώ το ελεκτικό συνέδριο για την λεπτομερή αξιολόγηση που δείχνει και τον τρόπο με τον οποίο θα υπερβούμε τα προβλήματα αυτά. Επίσης είμαστε ικανοποιημένοι με την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δέχεται όλες ε, τις συστάσεις. Όσον αφορά τις πληροφορίες ε, από ε, τις πληροφορίες που έχουμε λάβει, ε, θέλω να απευθύνω δύο ερωτήσει στην Κομισιόν. Όσον αφορά τη διευκόλυνση και τους πρόσφυγες στην Τουρκία, η Διοικητική Επιτροπή είναι έτοιμη, η Διεχειριστική Επιτροπή να υλοποιήσει τα διδάγματα που αναφέρονται στη διαδικασία ορισμού των βασικών προτεραιοτήτων για τη δεύτερη φάση της διευκόλυνσης. Και δεύτερον, πώς σκοπεύετε να βελτιώσετε την κατανομή της χρηματοδότησης ώστε να είναι αναλογική βάσει των αναγκών σε κάθε τομέα προτεραιότητας. Επίσης χρειάζονται κάποιες εξηγήσει όσον αφορά τη χρηματοδότηση που αναφέρθηκε. Η τουρκική κυβέρνηση, όπως φαίνεται, δεν λαμβάνει αυτά τα χρήματα ίδια. Τα χρήματα αυτά διέρχονται μέσω των 72 ή 74 έργων, δεν θυμάμαι σίγουρα πόσα είναι. Και αυτό χρειάζεται κάποια διευκρίνηση. Πρέπει να ενημερωθούν σχετικά οι ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ. Ναι, έχω γράψει και το δικό μου όνομα στο κατάλογο των ομιλητών. Θέλω να μου διευκρινίσετε κάποια άλλα πράγματα. Και η Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού, θυμάμαι, είχε μεταβεί εκεί και στον Καζιαντέπ και στα σύνορα με τη Συρία. Ασχοληθήκαμε εντατικά με το σύστημα υποστήριξης με μετρητά, με κάποιες κάρτες που τους δίνουν. Είναι το σημαντικότερο και το μεγαλύτερο από πλευράς χρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέει ότι με αυτή την κάρτα δεν μπορούν να κάνουν ανάληψη σε μετρητά. Όμω η έκθεση λέει ότι μπορούν. Ε, μπορούν ή δεν μπορούν τώρα. Ποιο είναι το σωστό. Και δεύτερη ερώτηση. Πώς είναι δυνατόν. Πώς είναι δυνατόν να σεμνινόμαστε ότι έχουμε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα χωρίς να ξέρουμε αν το πρόγραμμα έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Και βγαίνουμε και διαδιπανίζουμε σε όλο τον κόσμο ότι τι σπουδαίο πρόγραμμα έχουμε φτιάξει. Σε κάθε μία ομιλία μου ε, παρουσιάζω αυτό το πρόγραμμα. Και τώρα ε, θα ήθελα πραγματικά να μου πείτε αν κοροϊδεύω τον κόσμο. Ε, τώρα ποιος έχει το λόγο από τη Γενική Διεύθυνση την αρμόδια. Η κυρία Φεράνη, ο κύριος Δεμπράου από τη Γενική Διεύθυνση έχω για την ανθρωπιστική βοήθεια. Ποιος θέλει, ποια, όποια σειρά θέλετε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ από την ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ και μαζί με τον Γενικό Διευθυντή της ΓΑΜΑ ΕΚΟ έχουμε συνεργαστεί από την αρχή του σχηματισμού της διευκολύνσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις Επιτροπές του Κοινοβουλίου για την πρόσκληση και το Ελεκτικό Συνέδριο για την εξαιρετική συνεργασία και έκθεση. Όπως αναφέρθηκε, η Κομισιόν αποδέχεται όλες τις συστάσεις και αυτή τη στιγμή κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να τις υλοποιήσει. Και για την υλοποίηση των έργων και για το σχεδιασμό της δεύτερης φάσης της διευκόλυνσης του μέσου. Ένα στοιχείο για το οποίο πραγματικά ευχαριστούμε θερμά το ελεγκτικό συνέδριο είναι ότι συνυπολόγησε την περιπλοκότητα του πεδίου, του περιβάλλοντος, το οποίο τα κάναμε όλα αυτά. Γιατί πρέπει να μην ξεχνούμε ότι εδώ δεν μιλούμε για χρηματοδοτικό μέσο. Μιλούμε για πλατφόρμα συντονισμού που σχεδιάστηκε εν μέσω μεταναστευτικής κρίσης προκειμένου να δράσουμε ταχαίως και αποτελεσματικά για να δώσουμε βοήθεια στους πρόσφυγες αυτούς. Σε ένα πραγματικά πολύ δύσκολο για αυτούς πλαίσιο και επομένως αναγνωρίζουμε απολύτως τις συστάσεις για βελτίωση και αναγνωρίζουμε ότι δεν ήταν όλα τέλεια από την πρώτη μέρα. Να απαντήσω λοιπόν άμεσα στην ερώτησή σας έχει αντίκτυπο στο έδαφος αυτό το μέσο. Ναι, έχει. Αλλά πρέπει να δει κανεί ότι η έκθεση αυτή εξετάζει την περίοδο Μάρτιος 16, Μάρτιος 18. Η διευκόλυνση σχεδιάστηκε το Φεβρουάριο του 16, δηλαδή μιλούμε για την πρώτη, την πρώιμη φάση της υλοποίησης. Βλέπουμε αποτελέσματα, αλλά είναι μόνο 10 έργα που ελέγχθηκαν από τα 72 γιατί ήμασταν στις αρχικές φάσεις υλοποίησής τους και επομένως συν το χρόνο θα συλλέγουμε ακόμα περισσότερες ε, πληροφορίες και δεδομένα για τα παραδοτέα και την αποτελεσματικότητα των έργων. Επίσης, το πλαίσιο είναι πληρέστερο ώστε να έχουμε τα δεδομένα που χρειαζόμαστε για την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο της υλοποίησης των έργων. Τώρα, τι κάνουμε για να υλοποιήσουμε τις συστάσεις. Θα ξεκινήσω από τις τρεις βασικότερες για την αποτελεσματικότητα συνολικά και σημείωσα τα σχόλιά σας για τα, ο έμεσο κόστος. Εμείς υλοποιούμε εντός του νομικού πλαισίου τις σχέσεις μας, δηλαδή με τους εταίρους υλοποίησης και με αυτό που καλούμε φάφα με τους οργανισμούς των ΗΕ και τους άλλους διεθνείς οργανισμούς σε συνεχή διάλογο μαζί τους ώστε να κατεβάσουμε, να περιορίσουμε αυτά τα έμεσα κόστη. Επίσης δημοσιεύσαμε δύο διαγωνισμούς στην δεύτερη δέσμη καταβολής όπου έχουμε ορίσει το πλεονασματικό κόστος 4% επί τη βάση της εμπειρίας που είχαμε από την πρώτη καταβολή. Για το streamlining. Όπως είπα, ε, μιλούμε για μια πλατφόρμα συντονισμού μεταξύ υφισταμένων μέσων την ανθρωπιστική βοήθεια των Εθνών, διάφορα έργα προενταξιακής βοήθειας, κυρίως υπό τη δεύτερη δέσμη του και ταυτόχρονα είχαμε την επιθυμία ταχείας υλοποίησης του μέσου αυτού της διευκόλυνσης ώστε να έχουμε και bottom-up και top-down προσεγγίσεις. Όταν ξεκίνησαμε το Μάρτιο, δεν ξεκίνησαμε εν κενό, Από το 2011 είχαμε ελοποιήσει ήδη έργα 350 εκατομμύριων ευρώ στο πεδίο και επομένως ξεκινήσαμε ήδη πριν τη δημιουργία της διευκόλυνσης με τους εταίρους υλοποίησης που έχουμε στο έδαφος. Συνδυάσαμε λοιπόν μεταξύ έργων που ήταν έτοιμα προς υλοποίηση και σχεδιασμό μεγαλύτερων, μεγαλύτερης κλέμακας έργων. Και πολύ σημαντικό εξ αυτών είναι το ESSN και η συνεργασία που έχουμε με τα Υπουργεία υγεία και Παιδεία στην Τουρκία. Αυτά βεβαίως απαιτούσαν χρόνο και οι τοπικοί εταίροι ήταν έτοιμοι να μας βοηθήσουν με συμπληρωματικά έργα που ήμασταν έτοιμοι να στηρίξουμε. Επομένω, ναι, είχαμε διάφορους εταίρου είχαμε τα έμεσα ε, έργα σε συνεργασία με τα Υπουργεία και είχαμε και τα έργα υπό τα Ηνωμένα Έθνη και πολύ σημαντικό στοιχείο της έκθεσης του συνεδρίου είναι ότι εξασφαλίζουμε διαρκώς ότι αποφεύγουμε κάθε είδους επικάλυψη ώστε να έχουμε ένα μείγμα εργαλείων που δίδουν αποτελέσματα και που συμπληρώνουν το ένα το άλλο. Για τη βιωσιμότητα και τη μεταβατική περίοδο, τη μετάβαση, είναι από τους βασικότερους μοχλούς προγραμματισμούς την δεύτερη δέσμη καταβολής, την οποία υλοποιούμε αυτή τη στιγμή, τα δεύτερα τρία δισεκατομμύρια, η παρέμβαση μέσω της διευκόλυνσης δεν σταματάει βεβαίως όταν ολοκληρωθεί η ενωσιακή χρηματοδότηση. Συνεργαζόμαστε με τις τουρκικές αρχές κατά τρόπον ώστε να είναι βιώσιμα τα πράγματα αυτά και ανάλογα με τη φύση του καθενός να αναλάβει η τουρκική κυβέρνηση κάποια από αυτά όταν ολοκληρωθεί, όταν σταματήσει η διευκόλυνση. Αυτό είναι ιδιαίτερο σημαντικό για τις δύο βασικές προτεραιότητες υπό τη δεύτερη δέσμη και που όπως είπε το Ενακτικό Συνέδριο είχαν λιγότερη ενίσχυση στην πρώτη δέσμη. Ε, βοήθεια προς τους τοπικούς δήμους και προς την υποδομή. Και εδώ προσπαθούμε να πάμε από την ανθρωπιστική κατάσταση σε πιο βιώσιμες και ολοκληρωμένες προσεγγίσεις υπό τις οποίες ανοίγουμε την αγορά εργασίας και μια βιώσιμη διαβίωση, για να το πούμε έτσι, των ανθρώπων αυτών όσο καιρό βρίσκονται στο έδαφος της Τουρκίας. Και αφού ολοκληρωθεί, αφού θα έχει ολοκληρωθεί η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να απαντήσω στην κάτι για την διαχείριση της μετανάστευσης που είναι ένα από τα επιλέξιμα πεδία υπό τη διευκόλυνση. Στην πρώτη δέσμη την, χρησιμοποίησαμε για έκτακτες ανάγκες. 20 εκατομμύρια είχαμε για τα σκάφη περιπολίας που χρειαζόντουσαν τότε και άλλο ένα για τις επιστροφές προς την Τουρκία με τη βοήθεια του γενικού, της Γενικής Διεύθυνσης ε, Διαχείρισης Μετανάστευσης. Δεν το βλέπουμε όμως προτεραιότητα κλειδί συνολικά η διευκόλυνση, που είναι άμεση ενίσχυση στους ίδιους τους πρόσφυγες. Παρόλα αυτά, αυτές οι ρήτρες ήταν απαραίτητες, διότι ήμασταν σε ένα πλαίσιο γενικότερης διαπραγμάτευσης με τις τουρκικές αρχές για το προσφυγικό και ένα από τα στοιχεία του Μαρτίου του 16 της δήλωσης δηλαδή, ήταν αυτό. Και αφήσαμε στην δεύτερη δέσμη δυνητική ενίσχυση βοήθεια που δεν είχαμε σχεδιάσει εξ αρχής αναγκαστικά στο, στη χρηματοδότησή της γιατί εξαρτάται λίγο και από τις ροές, τις ροές. Θεωρούμε πάντως ότι τα μέσα προενταξιακής βοήθειας και η βοήθεια προς την Τουρκία θα πρέπει να είναι το προνόμιο της ενίσχυσης των, της διαχείρισης των συνόρων από πλευράς Τουρκίας και της διαχείρισης του μεταναστευτικού. Επομένως είναι ένα δίκτυο ασφαλείας, αλλά δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα του μέσου. Θα έδινα τώρα το λόγο στον Ζων Λουί για πιο λεπτομερή στοιχεία για τα ανθρωπιστικά έργα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ακούγεται ο μιλητής δυστυχώς χωρίς μικρόφωνο. Δυστυχώ δεν ακούγεται ο μιλητής, δεν ακούγεται το μικρόφωνο. Move. Just move to. Okay. Ευχαριστούμε και πάλι για την υποδοχή σας ε, σήμερα το μεσημέρι. Ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να εκφράσουμε την εκτίμησή μας για τη συμβολή του ελεγκτικού συνεδρίου στην υλοποίηση του ESSN. Πάλι εκτό μικροφώνου. Δεν λειτουργεί δυστυχώ το μικρόφωνο του ομιλητή. Αλλάξτε μικρόφωνο σας παρακαλώ. Let me try again. Ας ξαναπροσπαθήσω. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Οι δύο βασικές ερωτήσεις είχαν ως εξής. Η πρώτη αφορούσε την πρόσβαση στα δεδομένα και ε, το ρόλο των ΜΚΟ. Ο ρόλος των ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη σε κάθε διάλογο που έχουμε με τις ε, τουρκικές αρχές. Τους εξηγούμε σαφέστατα ότι είναι απολύτως αναγκαίος εταίρος για την υλοποίηση ορισμένων από τα έργα στο ανθρωπιστικό σκέλος του SSN, ειδικότερα όσον αφορά τα θέματα προστασίας. Θεωρητικά το κατανοούν, πιστεύω, αλλά εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. στις αρχές συνέβη το εξώς η εργατική νομοθεσία της Τουρκίας δεν είναι γνωστή σε όλου του εταίρου και έκαναν η ΜΚΟ κάποια λάθη. Εμεί βοηθήσαμε στο να διορθωθούν αυτά τα λάθη και προτείναμε επισταμένα στι τουρκικέ αρχέ να εξηγούν και να παρουσιάσουν καθαρά τι απαιτήσει του όσον αφορά τη λειτουργία των μη κυβερνητικών οργανώσεων με κάποιο είδου εγκύκλιο που θα μπορούσαν να διαθέσουν σε όλου ε, και την οποία όλοι θα μπορούν να λάβουν υπόψη και να την υλοποιήσουν. Υπήρξε μάλιστα και ένα σχέδιο τέτοια ε, εγκυκλίου που έδωσαν οι οργανισμοί των ΗΕ στι τουρκικέ αρχέ. Δυστυχώ οι τουρκικέ αρχέ δεν ακολούθησαν αυτή την προσέγγιση. Εξακολουθούν να ακολουθούν μια προσέγγιση αντόκα. Κάθε φορά που πρέπει να γίνει ανανέωση ε, της τη εγγραφή τη αδειοδότηση κάποια ΜΚΟ ή τη ε, ενό μέλου των μακροχρόνια αυτό δεν είναι βιώσιμο. Ο Επίτροπος Στυλιανίδης στην πρόσφατη επισκεπτή του στην Τουρκία το επανέλαβε στις 8 Ιανουαρίου. Και σίγουρα θα επανέλθουμε σε αυτό ε, με τους ε, Τούρκους συνομιλητές μας. Υπάρχει και σαφή σύσταση ε, που το υποστηρίζει αυτό από το ελεγκτικό συνέδριο και αυτό δείχνει πόσο πολλοί μπορούν να βοηθήσουν τέτοιου είδου συστάσει. Ακούστηκε μία ερώτηση για τους εταίρους μας. Πρέπει να τονίσω ότι Σύμφωνα με το είπε η Μίρια, στην πραγματικότητα όλοι μας υλοποιούμε τη διευκολύνση σύμφωνα με το δικό μας νομοθετικό πλαίσιο. Ο κανονισμός ανθρωπιστικής βοήθειας μας, δίνει, μας επιτρέπει να συνεργαζόμαστε με τρεις τύπους εταίρων. Ε, ΜΚΟ, με την οικογένεια του Ερυθρού Σταυρού και τους οργανισμούς των ΗΠΑ. Δεν χρηματοδοτούμε, ούτε έχουμε τέτοια άδεια ε, ευρωπαϊκούς οργανισμούς, ούτε κράτη το οποίο εξηγεί για ποιο λόγο εργαζόμαστε μέσω του WFP. Ε, γιατί η ερώτηση ήταν γιατί δεν εργάζεται απευθείας ε, με τον ε, τον Σταυρό της Τουρκίας. Ε, όπως φαίνεται θα χρειαστεί χρόνο μέχρι να εγγραφεί ως εταίρος με την Εμισέλινο. με την Ερυθρέα Μισελέα της Τουρκίας ε, υπήρξε μια συμφωνία για να καλύψει το κόστος της ε, συμβολής ε, στη δράση αυτή. Συγγνώμη, αναφερόταν στο Παγκόσμιο Επιστημιστικό Πρόγραμμα ο ομιλητής. Όσον αφορά την πρόσβαση στα δεδομένα των δικαιούχων, αναφέρθηκε ότι αυτό αποτελεί συνέπεια τη νομοθεσία προστασία δεδομένων τη Τουρκία. Και πρέπει να πω ότι αυτή η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων τη Τουρκία βασίζεται σε ένα σύστημα κοντινό στο δικό μα. Αφορά τη μεταφορά δεδομένων εκτός Τουρκίας σε μη τουρκικούς οργανισμούς. Οπότε πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή. Ε, αν προσπαθούμε να αγγίξουμε αυτό το ζήτημα υπάρχει ένα αυστηρό σύστημα ταυτοποίηση, όπω έχει ζητηθεί, αλλά χρειάζεται και κάποια διευκρίνηση, διότι και εμεί πιστεύουμε ότι μπορούμε να είμαστε καθυσυχασμένοι αυτή τη στιγμή, παρότι θα συνεχιστούν οι συζητήσει. Πώ φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση. Υπάρχει μια διμερή συμφωνία, όπω είπα νωρίτερα, μεταξύ τη Τουρκική μισελίνου και των διαφόρων υπουργείων που επιτρέπει την ανταλλαγή μεταξύ αυτών των υπουργείων και τη Τουρκική ημισελήνου για τα εξή ε, προσωπικά δεδομένα. Όνομα, επώνυμα, ε, αριθμό ταυτότητας, ε, γειτονιά κατοικία και τηλέφωνα. Αυτές οι πληροφορίες μετατρέπονται από την GRC μέσω ενό αλγορίθμου που παρέχει για κάθε δικαιούχο, κάθε νοικοκυριό, έναν συνολικό αριθμό ταυτότητας και έναν ανώνυμο αριθμό ταυτότητας ε, στο WFP. Το Παγκόσμιο Επιστημιστικό Πρόγραμμα WFP επίσης έχει πρόσβαση στον αριθμό πελάτη. Ταυτοποίησης πελάτη. Υπάρχει λοιπόν κάποια ασθενή σύνδεση μεταξύ των ανώνυμων δεδομένων που έχει το WFP και τα μη επεξεργασμένα βιογραφικά δεδομένα που έχει στα χέρια του η τουρκική συστηματικά ελέγχονται αυτές οι πληροφορίες και συγκρίνονται οι πληροφορίες αυτές μεταξύ των δύο οργανισμών και ειδικότερα όταν εφαρμόζει την διαδικασία επαλήθευσης ε, το WFP. Μέχρι στιγμής δεν έχει παρατηρηθεί κανένα πρόβλημα, καμία έλλειψη. Καμιά φορά υπάρχει ασυμφωνία πληροφοριών, αλλά αυτές ε, διορθώνονται ικανοποιητικά. Παρ' όλα αυτά δεν πάβουν να είναι διαμεσολαβητές. Και ε, στην τελευταία επισκέψη του Επιτρόπου Στυλιανίδη στην Τουρκία είπαμε ότι θα συνεχίσουμε να διερευνούμε λύσεις σε τεχνικό επίπεδο ορισμένες από τις οποίες μπορεί να έχουν ως εξή να δούμε κατά πόσο μπορούν να υπάρξουν εξαιρέσει που να επιτρέπονται από την τουρκική νομοθεσία προστασία δεδομένων. Αυτό μπορούμε να το μελετήσουμε επίση. Μπορεί να προκύψει και κάποια άλλη λύση να επενδύσουμε, να συμφωνήσουμε να επενδύσουμε σε ένα έμπιστο τρίτο μέρος το οποίο θα παρακολουθεί αυτή τη διμερή σχέση μεταξύ όσων λειτουργούν το ESSN, δηλαδή η Ερθρά, η Μισέλινος και WFP και οποιοδήποτε άλλοι θα το χρησιμοποιούν στο μέλλον. Οπότε οι προσπάθειες είναι να εξελίξει και σαφής ε, σύσταση όπως είπα, ε, όπως αυτή που έχουμε από το ελεκτικό συνεδρίο θα μας βοηθήσει να τροφοδοτήσουμε αυτό το διάλογο με τις τουρκικές αρχές. Ζητώ συγγνώμη, βλέπω ότι μίλησα παραπάνω ώρα από ό,τι μου επιτρέψατε, αλλά ήθελα να καλύψω τα βασικά ζητήματα. Για μένα δεν μακρηγορήσατε. Καθόλου. Δηλαδή, τώρα εσείς μπορεί να εγγυηθείτε ότι τα χρήματα ε, φτάνει στους δικαιούχους που πρέπει, ε, δηλαδή στους πρόσφυγες με αυτές τις κάρτες, παρόλο που το ελεγκτικό συνέδριο δεν μπορεί να παρακολουθήσει τη διαδρομή του χρήματος από την εκταμείευση μέχρι τη τελική του καταβολή. Να διευκρινίσω κάτι. Ε, η τουρκική ερυθρά ε, πληρώνει, όχι το τουρκικό κράτος. Ποιος δίνει τα λεφτά στον κόσμο. Η, τουρκική ερυθρά Έλληνος Ναι, ακριβώς. Απολύτως. Πρόεδρε, γνωρίζετε κι εσείς πώς λειτουργούμε. Τα χρήματα αυτά δεν πηγαίνουν στο τουρκικό κράτος. Δεν συνεργαζόμαστε με το τουρκικό κράτος, το οποίο κατά τα άλλα ε, δεν διευκόλυνε την κατάσταση γιατί είχε την αιμονή ε, να περνάνε τα χρήματα μέσω του τουρκικού κράτους. Εμείς ε, εκτελούμε το ανθρωπιστικό σκέλος ε, της βοήθειας ανάλογα με τον αντίστοιχο κανονισμό που δεν συνεργαζόμαστε με κρατικές ή κρατικού τύπου οργανώσεις, αλλά με την τουρκική ερυθρά ή μισέλινο. Συγγνώμη, ξέχασα να σας απαντήσω για τις κάρτες. Δεν είναι η κάρτα που μπορεί να ε, ε, επιτρέπει ε, να γίνονται αναλήψεις μετρητών από το ATM. Είναι ένα σύστημα με voucher, με δελτία δηλαδή, που παίρνουν ας πούμε σε είδος κάποια βοήθεια όπως είναι τρόφιμα και πληρώνουμε την κάρτα. Λέτε ότι δεν έχετε επιφυλάξει λοιπόν ότι τα χρήματα ε, δεν φτάνει ε, στους δικαιούχους, ε, σε αυτούς που, για τους οποίους έχουν σχεδιαστεί. Ναι, ναι, εμείς πιστεύουμε ότι το σύστημα προς το παρόν λειτουργεί και είναι απολύτως οχυρωμένο. Βέβαια, συμφωνούμε με το ελεκτικό συνέδριο ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε πιο εύκολα και πιο απλά όλα αυτά τα πράγματα χωρίς ε, διάμεσους, αλλά χρησιμοποιούμε τις τους δύο διάβλους που σας ανέφερα προηγουμένως. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γιάκοψεν, παρακαλώ. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να αναφερθώ σε κάποιες από τις ερωτήσεις που έγιναν για το διοικητικό κόστος και το επιπλέον κόστος. Το 7% που αναφέραμε είναι τα χρήματα που θα καταβληθούν. Δεν υπάρχει άλλο πρόσθετο πάνω σε αυτά. Είναι το 7% που αναφέρεται και στη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τα, τη διαχείριση των, της μετανάστευσης, τα δύο έργα που αναφέρατε δεν ήταν μεταξύ αυτών που ελέγξαμε, αλλά μπορούσαμε να δούμε ότι η Επιτροπή Καθοδήγησης αποφάσισε να μην συνεχίσει με πόρους στο πεδίο αυτό, γιατί στον έλεγχο είδαμε ότι δεν ήταν αυτό που είχε συσταθεί ως στόχος του όλου μέσου της όλης διευκόλυνση. Επομένως δεν έχουμε δεδομένα για εκείνα τα δύο συγκεκριμένα έργα. Έγιναν επίσης κάποιες αναφορές ε, στην, ε, στα εκπαιδευτικά και την αξιολόγησή μας των διαφόρων έργων. Στο παράδειγμα 3B έχουμε μία αξιολόγηση με χρώματα, το πράσινο είναι αυτό που τα πάει πολύ καλά, το κίτρινο έτσι και έτσι και τα κόκκινα αυτά που δεν λειτουργούν καλά. Και επί τη βάση, μάλλον η συνολική εικόνα είναι ε, μία ανάμεικτη αξιολόγηση για το πώς βλέπουμε τα διάφορα έργα. Ε, μας ρωτήσατε και για τις εντυπώσεις μας για τα έργα εκπαίδευσης. Στο παράδειγμα 7 επίσης είχαμε κάποια παραδείγματα των διαφόρων εκπαιδευτικών έργων με ποιος είναι χορηγός ποιας πρωτοβουλίας, μαθήματα τουρκικής γλώσσας, ε, κατάρτιση, είναι ανάμειξη διαφόρων χορηγών και διαφόρων εργών που καλύπτουν τον τομέα της παιδείας, αλλά στο παράδειγμα 7 μπορείτε να δείτε όλες τις δραστηριότητε και είναι αρκετές που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της ε, παιδείας. Έχουμε και τα έργα με τις ε, προϋποθέσεις για μεταφορά χρημάτων ρευστού για τα προγράμματα επίσημης εκπαίδευσης ώστε τα παιδιά των προσφύγων να επιλέξουν την παιδεία που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν. Και τέλος, ε, για την ερώτηση του κατά πόσον έχει κανείς λαμβάνει ρευστό στο χέρι, πρόκειται για χρεωστική κάρτα με την οποία μπορεί κανείς να λάβει χρήματα από το ATM ή να πληρώσει στα καταστήματα. Είναι λοιπόν δυνατόν να λάβει κανείς τελικώς χρήματα ρευστό στο χέρι. Αυτά. Ευχαριστώ. Σύντομα κυρία Κινίτση για να κλείσετε παρακαλώ. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφου που παρενέβησαν και την κυρία Γιάκοψεν και πάλι, όπω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι προέκυψε από τη συζήτηση ότι πραγματικά συζητούμε για ένα πολύ σημαντικό μέσο και σε σχέση με τις ανθρωπιστικές του στοχεύσεις που πιστεύω συμφωνούμε όλοι. Αλλά ακριβώς γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε έναν προσεκτικό έλεγχο για την εξέλιξη των έργων, για τη χρησιμοποίηση των κονδυλίων χρηματοδότησης και όχι μόνο για τις εκροές αλλά και για την επίτευξη των στόχων που χρηματοδοτούμε. Ε, μου φάνηκε αυτό πολύ σημαντικό όταν ελέγχθη και από την Κομισιόν και πάλι από την κυρία Γιάκοψεν ε, για το είδος του ελέγχου που διεξάγεται και κατά τη γνώμη μας πρέπει να είναι κάτι στο οποίο πρέπει να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο και σε πολιτικό επίπεδο με τις τουρκικές αρχές. Είναι πολύ σημαντική επίσης η ενίσχυση προς τις ΜΚΟ, το είπαμε, διότι ακριβώς το πεδίο αυτό ε, κάνουν πολύ σημαντική δουλειά και πρέπει να πω επίσης ότι θα συμφωνούσα με τα όσα είπε η Κομισιόν σχετικά με τις ε, λεπτομέρειες, της διευθετήσεις της δεύτερης δέσμης χρηματοδότησης για την βιωσιμότητα της δεύτερης φάσης του προγράμματος ακριβώς προκειμένου να δοθεί μια συνέχεια με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα μπορέσει να παράσχει αποτελεσματικότητα σε όλα τα έργα που θα έχουν κινήσει, ακόμα και όταν θα τερματιστεί η χρηματοδότηση η ενωσιακή. Νομίζω ότι και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπό το συνολικό οπτικό Και θα ήθελα λοιπόν να κλείσω ευχαριστώντα και πάλι όλου για τη συνεισφορά του και επαναλαμβάνοντα ότι το μέσο είναι αποτελεσματικό αλλά ακριβώ γι' αυτό και επειδή παρέχει βοήθεια χρειάζεται προσεκτικό έλεγχο. σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Και εγώ σε ευχαριστώ. Είπαμε στο σημείο 11. Συνεχίζουμε με την κυρία Γιάκοψεν ε, για το καταπιστευματικό ταμείο για την Αφρική. Να μην σα πω ότι έχουμε και μισή ώρα καθυστέρηση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω την ειδική έκθεση για το Πιστευματικό Ταμείο Εκτακτής Ανάγκης Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αφρική. Όπως γνωρίζετε από το 2013 ο Δημοσιονομικός Κανονισμός επέτρεψε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργεί καταπιστευματικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αυτά ε, συναπαρτίζονται από κονδύλια του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού ή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης μαζί με άλλους δωρητές, έναν ιδίων, συμπεριλαμβανομένων και ε, των κρατών μελών ή άλλων κρατών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ταμείο αυτό για την Αφρική στόχο έχει να σφυρλατήσει την σταθερότητα και να βοηθήσει να γίνεται καλύτερα διαχείριση της μετανάστευσης αντιμετωπίζοντας τη ρίζα ε, του κακού ε, της αποψήλωση των δασών, τη αναγκαστική μετανάστευση και τη παράνομη μετανάστευση. Το Νοέμβριο του 2015 έθηκε ε, η πρώτη, τα πρώτα θεμέλια. Ε, τώρα είναι η τέταρτη προσπάθεια υποστηρίζουμε ε, σε τρεις περιφέρειες 26 χώρες. Οι τρεις περιφέρειες ονομάζονται ε, θηρίδες ή παράθυρα, ε, Σαχέλ και Λίμνη Τσάλτ, Κέρας της Αφρικής και Βόρεια Αφρική είναι οι τρεις περιφέρειες. Από το 2015 μέχρι τα τέλη του 2020 αναμένεται να λειτουργεί αυτό το καταπιστευματικό ταμείο και τέλος Αυγούστου του 2018 οι συνεισφορές ήταν πάνω από 4 δις ευρώ το 89% του συνόλου των συνεισφορών είναι μεταβιβάσεις από το Ευρωπαϊκό Προπολογισμό και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Στόχος μας ε, στον έλεγχο που κάναμε ήταν να δούμε αν ήταν καλά σχεδιασμένο και αν εφαρμόζεται καλά αυτό το καταπιστευματικό ταμείο. Ε, πρώτα εξετάσαμε το σχεδιασμό, ε, του στόχου, την ανάλυση των αναγκών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη χρηματοδότηση. Στη συνέχεια εξετάσαμε ειδικά στοιχεία και πτυχές από την υλοποίηση εκτέλεση του Ταμείου, ε, διαδικασίες επιλογής για τα έργα, σύστημα παρακολούθησης και αποτέλεσμα που ρίχαν τα έργα τα οποία ελέγξαμε. Επίσης κάναμε και επιτόπιους ελέγχους με επίσκεψη στον Ήγυρα και την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωση στη Λιβύη και εξετάσαμε 20 προγράμματα που τρέχουν στις δύο αυτές χώρες. Και τι διαπιστώσαμε. Καταλήξαμε ότι το μέσο αυτό είναι ένα ευέλικτο εργαλείο, αλλά επειδή είναι πρωτοφανείς οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει, ο σχεδιασμός του θα έπρεπε να ήταν πιο στοχευμένος από την αρχή. Ένας από τους ευρύ, μάλλον οι ευρύ στόχοι που έχει επιτρέπουν ευελιξία, αλλά οι στρατηγικές είναι μάλλον κατακαιρματισμένες, δεν είναι αρκετά εστιασμένες για να κατευθύνουμε τις δράσεις και να μετράμε τον αντίκτυπο και στις τρεις περιφέρειες αυτές τις ρίδες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει κάνει μια συνολική αξιολόγηση των αναγκών που πρέπει να καλυφθούν, ούτε των μέσων που έχει στη διάθεσή της. Η στρατηγική καθοδήγηση που γίνεται προς τους διαχειριστές ε, των τριών θηρίδων δεν ήταν αρκετά ε, ειδικοί. Όλοι ε, και οι στόχοι δεν ήταν ποσοτικοποιημένοι. Όπως δεν έχει οριστεί η κρίσιμη μάζα χρηματοδότησης. Επίσης βρήκαμε ότι η συγκέντρωση των πόρων και των δυνατοτήτων δεν γίνεται με τρόπο πάντα αποτελεσματικό ούτε συστηματικό. Επίσης, δεν είχαμε και μηχανισμό για την εξαγωγή διδαγμάτων. Επίσης είδαμε ότι η διαδικασία επιλογής των ε, έργων διαφέρει από περιφέρεια σε περιφέρεια. Δεν βρήκαμε κανένα έγγραφο ε, με συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιολόγηση ε, των έργων. Και ξέρουμε ότι η έλλειψη τέτοιων σαφών κριτηρίων είναι κάτι το οποίο έχουν υποδείξει και κάποια κράτη-μέλη αρκετά. Ωστόσο, μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι δεν υπάρχει ανάγκη να τα διευκρινίσει. Το συγκριτικό πλεονέκτημα ε, γιατί είναι ε, πιο επωφελές ε, και πιο συμφέρον να χρηματοδοτούνται κάποια έργα από το καταπιστευματικό ταμείο. Αυτό δεν έχει εξηγηθεί επαρκώς. Και σε σύγκριση με παραδοσιακά εργαλεία, ε, στη φάση της αρχικής χρηματοδότησης και λειτουργίας, πραγματικά είναι ταχύτερο για τις προκαταβολές και για να τεθούν σε λειτουργία κάποιες διαδικασίες. Ωστόσο, τα έργα αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα και δυσκολίες, ε, όπως και με παραδοσιακά μέσα χρηματοδότησης που καθυστερούν την υλοποίησή τους ενώ ε, το καταπιστευματικό ταμείο ε, ε, πρέπει να απαντήσει σε μια έκτακτη ανάγκη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει προβλέψει έκτακτα έργα για να διευκολύνουν και μέσα την εργασία των εταίρων για να μπορούν να λειτουργούν και να αρχίζουν νωρίτερα. Υπάρχει ένα κοινό σύστημα ελέγχου, αλλά δεν έχει ακόμα τεθεί σε λειτουργία. Και οι τρεις περιφέρειες μέχρι τώρα χρησιμοποιούν διαφορετικά συστήματα για να συλλέγουν ε, πληροφορίες για τον προβλογισμό, να κάνουν τον έλεγχο και την παρακολούθηση και την αξιολόγηση. Ε, και οι στόχοι των έργων δεν ήταν πάντα ευφυείς, ούτε οι δείκτες που χρησιμοποιούνται ε, για να μετρούν την απόδοση εύστοχοι. μπορεί με να έχει μειωθεί ο αριθμός των παράτυπων μεταναστών που περνούν από την Αφρική στην Ευρώπη. Ε, δεν ξέρουμε με ποσοτικούς όρους πόσο έχει συνεισφέρει σε αυτό το καταπιστευαντικό ταμείο. Τώρα έχουν αρχίσει να φαίνονται τα πρώτα αποτελέσματα από τα έργα που έχουν στηθεί. Ένα έργο ε, είχε στόχο να δώσει συνθήκες ε, διαβίωσης ε, αξιοπρεπής. Το 2017 πάνω από 9.000 πρόσφυγες στον Ήγηρα συμμετείχαν. Ε, αλλού 19 διεθνή δίκτυα διακίνησης διαλύθηκαν ε, χάρη στις κοινέ έρευνες αστυνομικέ και άλλων ερευνητικών αρχών το 2017 στον Ήγηρα πάλι. Στη Λιβύη υποστηρίχθηκαν 4.700 πρόσφυγες για ε, ε, ε, επιστροφή τους εθελούσια, ενώ περίπου 20.000 άλλοι υποστηρίχθηκαν. Τι λέμε στις συστάσεις μας. Τέσσερις συστάσεις έχουμε κάνει για να βελτιωθεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση και η εκτέλεση αυτού του καταπιστηματικού ταμείου για την Αφρική. Θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να βελτιώσει την ποιότητα των στόχων και των προτεραιοτήτων, έτσι ώστε το Ταμείο να έχει συγκεκριμένου στόχου και πιο εφικτού, να αναθεωρήσουν τη διαδικασία επιλογή των έργων για να είναι πιο συνεκτική και πιο διαφανής. Θα πρέπει να πάρουν μέτρα για να επιτεχυνθεί η υλοποίηση και τέλος να βελτιώσει τον έλεγχο και την παρακολούθηση του καταπιστευματικού ταμείου. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επικοδομητική της συνεργασία δέχθηκε τις περισσότερες στάσεις μας, αλλά κυρίως εκείνες που στοχεύουν στο να ε, διευκρινίζονται τα κριτήρια για την επιλεξιμότητα των έργων ε, είναι κάτι το οποίο δεν δέχτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ και περιμένω τα σχόλιά σας. Η, η συγγητριά μας η κυρία Γιάλα Σέντερ. ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν λειτουργεί το... το... Συγγνώμη, δεν σας έδωσα το λόγο, λέει η Πρόεδρος. Δεν είναι η δική σας σειρά. Πρώτα η συγγήτρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα σας ήμουν ευγνώμων καμιά φορά να κοιτάει και προς τα δω η γραμματεία, γιατί σε λίγο θα αρχίσω να χτυπάω παλαμάκια για να με δείτε, γιατί είχα και για την Τουρκία κάποιες ερωτήσεις, αλλά θα τις κάνω στις τροπολογίες μου. Τι να κάνω. Ευχαριστώ την κυρία Γιάκοψεν για την έκθεση αυτή και την παρουσίαση της ειδική έκθεσης. Είναι πολύ σημαντική γιατί βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, καθότι από το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το Ταμείο για την Ανάπτυξη το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη θα είναι ενταγμένο στον προπολογισμό. Και θα έχουμε και μια δυνατότητα ελέγχου, που ήταν και μια ερώτηση προς την κυρία Γιάκοψεν που θα είχα. Τι θα γίνει τώρα και πώς θα μπορούσαμε καλύτερα να ελέγχουμε αυτό το καταπίστευμα στο βαθμό που πολλά από τα χρήματα, τα ευρωπαϊκά, προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, που ήταν εκτός προϋπολογισμού μέχρι τώρα. Άρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ε, όπου πολλά από τα προβλήματα που βλέπουμε και που γνώρισαν σφοδρή κριτική ήταν ο τρόπος με τον οποίο συνεργάζεται με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αναπτυξιακή βοήθεια. Ότι μήπως θα μπορούσαμε να το είχαμε σχεδιάσει διαφορετικά. Σας ευχαριστώ για αυτά που είπατε. Αλλά υπάρχει κάτι που δεν βρίσκω εγώ στις απαντήσεις. Ξέρετε ότι υπήρξε μια σφοδρή αντίδραση να μην αλλάξουν οι στόχοι. Οι οποίοι ε, αυτοί οι στόχοι δεν είναι απλώς που αφορούν μια στρατηγική της επταετούς προγραμματικής περίοδου, αλλά ε, είναι και απορρέων από την ίδια τη συνθήκη. Τι σημαίνει αναπτυξιακή βοήθεια, βοήθεια να αναπτύσσονται οι χώρες που βρίσκονται σε μια κατάσταση φτώχειας, υπανάπτυξης, με μεγάλες ελλείψεις, ε, με λίγες αντιστάσεις απέναντι στην κλιματική αλλαγή κτλ. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι ε, ένα ταμείο έκτακτης ανάγκης, όπως είναι αυτό το καταπίστευμα, που έρχεται να απαντήσει ε, σε μια τραγωδία της τραγωδία μετανάστευσης, γιατί είναι τραγωδία και από τη σκοπιά της εκμετάλλευσης για του διακινητές, εκεί που πουλάνε ανθρώπους, οι δουλέμποροι στο Σαχέλ και σε όλα αυτά τα εδάφη και προς την Κεντρική και τη Δυτική Αφρική. Είδαμε ότι η οδός ε, μέσω της Τουρκίας κλείνει κατά κάποιο τρόπο και το συζητήσαμε και στο προηγούμενο θέμα και τώρα στρέφονται προς την άλλη πλευρά. Βλέπουμε να πνίγονται μετανάστες ε, στη Μεσόγειο. Ε, τα γνωρίζουμε όλα αυτά τα τραγικά. Λοιπόν, κυρία Γιάκοψεν, για ποιο λόγο η πρώτη σας σύσταση δεν ήταν αυτή. Ένα τέτοιο καταπιστευματικό ταμείο πώς αλλάζει ε, όταν αλλάζει η πηγή της χρηματοδότησης. Ξεφεύγουμε δηλαδή από την πάγια αναπτυξιακή βοήθεια και περνάμε προς την καταπολέμηση των αιτίων της μετανάστευσης, γιατί ξέρουμε ότι συνδέεται και η επανάπτυξη με τη μετανάστευση. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ε, κοντά, αλλά δεν έχουν τις ίδιες αιτίε. Και για τα υπόλοιπα στοιχεία, ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δέχτηκε τις συστάσεις ως προς την ιδιαιτερότητα των στόχων. Καταλαβαίνω και γιατί χώρες μιλάμε. Στη Λιβύη δεν μπορείς καν να πάει ε, το ελεγκτικό συνέδριο. Εμεί πήγαμε με μία ε, αποστολή πάρα πολύ δύσκολα. Δεν είναι μέρος η Λιβύη που να μπορείς να πας εκεί να ελέγξεις τις πληρωμές, αλλά μπορείς να ελέγξεις μέσω διεθνών οργανισμών ποιες είναι οι δυσκολίες εκτέλεσης των προγραμμάτων. και τα αποτελέσματα δεν είναι ποτέ επίγοντα έκτακτα ή βράχη είναι μέσο μακροπρόθεσμα. Ευχαριστώ λοιπόν και θα δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και να βεβαιωνόμαστε στο μέλλον για την εκτέλεση, να εξακριβώνουμε πώς εκτελούνται, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και το έκτακτο και το ευέλικτο, αλλά υπάρχουν και άλλες επιπτώσεις από όλα αυτά, πιο μακροπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες, που δείχνει ότι χρειάζονται και άλλες πολιτικές με περισσότερη πρόληψη. Και η ε, αδελφή η επιτροπή μας στο Bundestag θα ήξερε αυτά από το 2000 2000. Και εμεί αργήσαμε μέχρι το 2014, μέχρι το 2016 για να ξεκινήσει. Αλλά πρόβλημα έχουμε, αλλά το πρόβλημα δεν είναι στην Αφρική, είναι εδώ. Στην Αφρική έχουν άλλα προβλήματα. Εμείς κάναμε 15 χρόνια να το καταλάβουμε αυτό που συμβαίνει, για να αντιδράσουμε. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος Μακάλιστερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσει προς την κυρία Γιάκοψον. Η πρώτη έχει ως εξής. Ίσως να το γνωρίζετε, αλλά αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή ΑΦΕΤ συζητάμε δύο εκθέσεις για ο μέλλον της προενταξιακής βοήθειας και για την διεθνή ε, συνεργασία για το καταπίστευμα για την Αφρική αναφέρατε ότι η διακυβέρνηση γίνεται από την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη κυρίως και ότι δεν παίζει ρόλο ιδιαίτερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπορείτε να βελτι... Μπορεί να βελτιωθεί αυτό, θεωρείτε. Δεύτερη ερώτηση, μπορούμε να μάθουμε τίποτα από την εμπειρία του καταπιστεύματος για την Αφρική, για τα μελλοντικά καταπιστεύματα γενικότερα. Η κυρία Μακέβαν. Πρόεδρε, και εγώ είχα την ίδια ερώτηση, αλλά και σε σχέση με τα όσα είπε η κυρία Αγιάλα. Υπό τους κανόνες της σύστασης του καταπιστεύματος και υπό το χρηματοδοτικό κανονισμό, θα πρέπει τα κονδύλια να ευθυγραμμίζονται με τους στόχους των αναπτυξιακών πόρων από τους οποίους προέρχεται Είπατε ότι οι στόχοι ήταν σαφείς, αναλύσατε κατά πόσον τα κονδύλια, οι πόροι χρησιμοποιήθηκαν υπό τον αρχικό του σχεδιασμό. Επίσης λέτε ότι το ETE συνεισφέρει στη μείωση των παράνομων μεταναστών που κινούνται προς την Ευρώπη. Αυτό πώς το προσμετρήσατε, με ποιο τρόπο. Η κυρία Γκλαμπάγιοβα, ευχαριστώ πρόεδρε. Όπως και στο προηγούμενο σημείο και εδώ, θα χρησιμοποιήσω τον τίτλο της έκθεσης για να συνοψίσω. Το καταπίστευμα εκτάκτου ανάγκης είναι ευέλικτο, αλλά του λείπει λίγη εστίαση. Το ελεκτικό συνέδριο λέγει, καταρχάς μάλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει το καταπίστευμα ως κάτι που σχεδιάστηκε από τις ανάγκες που προκύπτουν από τις προκλήσεις και τις περίπλοκες ε, ε, τα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε. Αλλά και υπό τη ευρύτατο αυτό πεδίο θα πρέπει να έχουμε μια εστίαση, μια κατεύθυνση δηλαδή, ώστε να χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτή η εστίαση πώς ορίζεται καλύτερα. Εσείς τι θα προτείνατε. Επίσης λέγει το συνέδριο ότι ο στόχος και η παρακολούθησή τους, η παρακολούθηση των στόχων μάλλον, δεν ήταν πάντα ευφιέστατος. Τα μέτρα που λαμβάνονται ή που πρόκειται να ληφθούν θα επηρεάσουν τις τρέχουσες επιχειρήσεις. Δηλαδή αυτές που ήδη είναι σε λειτουργία θα έχουν έναν αντίκτυπο από αυτό. Συνάδελφος Στάς, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να συνεχίσω ε, ε, από αυτά που είπε η κυρία Μακάβαν. θα εχουν εναν αντικτυπο απο αυτο συνεδευος στας Γιάκοψεν, είπατε ότι το 89% των ε, χρημάτων προέρχονται από το Ταμείο Ανάπτυξη και τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Είναι αναπτυξιακά κονδύλια. Η Oxfam και η Concord, που είναι ο κεντρικός φορέας, υπολόγισε ότι το 22% πηγαίνει στην παρακολούθηση και φύλαξη των συνόρων, 15% στην ασφάλεια και καταπολέμηση βίου εξτρεμισμού από τα λεφτά τα ανθρωπιστικά. Λοιπόν, εγώ είμαι υπέρ. Καλό είναι ε, να γίνεται, αλλά πρέπει να παίρνουμε τα λεφτά από την ανθρωπιστική βοήθεια. Τα χρήματα της ανθρωπιστικής βοήθειας θα πρέπει να καταπολεμούν τη φτώχεια, την ανισότητα και να καλύπτουν τις ανάγκες των ανθρώπων για ανάπτυξη. Αυτό το έχετε μελετήσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει απάντηση σε αυτό. Δεύτερη ερώτηση. Μια άλλη κριτική της Oxfam και Concord είναι ότι όλο το καταπίστευμα για την Αφρική παραθέτω, με, λειτουργεί με τρόπο, με λήψη απόφασης και πάρα πολύ συγκεντρωτική και καθοδηγούμενη, με πάρα πολύ μικρή συμμετοχή και λόγω των τοπικών ΜΚΟ και των τοπικών αρχών. Όποιος έχει δουλέψει με την αναπτυξιακή βοήθεια ξέρει ότι αν δεν συμμετέχει ο κόσμος εκεί, αν δεν έχει λόγο για την απόφαση των έργων που επιλέγονται, στο Δίνεκε, τα χρήματα δεν πιάνουν τόπο και δεν έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό το έχετε μελετήσει. Η κυρία Γιάλα και πάλι σύντομα όμως, ναι. Θέλω να απαντήσω στον κύριο Μακάλιστερ ότι από το 2017 το Κοινοβούλιο έχει το καθεστώς του παρατηρητού σε αυτό ε, το καταπιστευματικό ταμείο. Δεν ξέρω ποιος εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο εκεί, πάντως το ζήτησε το Κοινοβούλιο και παρουσία έχουμε. Τώρα δεν ξέρω ποιος συμμετέχει εξ ονόματος του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ταμείο αυτό. Από τη Γενική Διεύθυνση ε, ΔΕΦΚΟ, ο κύριος Τόσπο και από την DGNIR ο άλλος συνάδελφος, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη που έκοψα κάποιον, δεν ήταν πρόθεσή μου. Είμαστε ικανοποιημένοι με την ειδική έκθεση για το ειδικό καταπίστευμα για την Αφρική. Συμφωνώ, ο διάλογος με το Αναλυτικό Συνέδριο υπήρξε επικοδομητικός και με, το ίδιο και με πολλούς ενδιαφορομένους κατά την υλοποίηση και πράγματι η έκθεση βοηθά ήδη σημαντικά στη βελτίωση ορισμένων πτυχών του καταπιστευματικού ταμείου. Ωστόσο, θα ήθελα να επενθυμίσω την κατάσταση που αντιμετώπισε το 2015 η Κομισιόν, όταν ξέσπασε η μεταναστευτική κρίση. Το πόσο επίγον ήταν να υποστηρίξει ε, να δράσει υποστηρικτικά η ευρωπαϊκή πλευρά. Φυσικά, εκ των υστέρων μπορεί να λέμε ναι, θα μπορούσαμε να είμαστε πιο εστιασμένοι στην αρχή, αλλά θυμηθείτε πόσο Επίγον ήταν το ζήτημα πολιτικά και απαιτούσε να αντιδράσουμε γρήγορα. Επίση, καλό θα ήταν να πούμε και αναγνωρίστε στην εκθέση, δεν αναφέρθηκε εδώ, ότι βαθμιά αυξήσαμε τη στρατηγική εστίαση. Από τις αρχές του 2017 είχαμε τακτικές συζητήσεις με το Συμβούλιο εκεί που καθίσει σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και είπα, μιλήσαμε για τη στρατηγική εστίαση που θα επιθυμούσαμε. Τα κράτη-μέλη δεν συμφωνούσαν για πάντα. Άλλοι θέλαμε να εστιαστούμε περισσότερο στην ανάπτυξη, άλλοι περισσότερο στη μετανάστευση. Χαιρόμαστε που το συνέδριο αναγνωρίζει το καταπιστευματικό ταμείο ως εργαλείο που βοηθά υποστήριξη των εταίρων σε πολλούς τομείς, πρόσβαση στην υγεία, παιδεία, ασφάλεια, βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργία οικονομικών ε, και επαγγελματικών ευκαιριών για ευάλωτες ομάδες όπως πρόσφυγες και εκτοπισμένους. Προφανώς σημειώνουμε και τις τέσσερις ε, συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Όπως προκύπτουν από την έκθεση, ήδη υλοποιούμε τις περισσότερες συστάσεις, αλλά υπάρχει μία που δεν δεχόμαστε. Αυτή αφορά τα κριτήρια επιλογής για, την, για τα έργα, γιατί δεν είναι πρόσκληση για συμμετοχή σε διαγωνισμό το καταπιστευματικό ταμείο. Ε, βρισκόμαστε σε διαβούλευση με του τοπικού ενδιαφερομένου, με τι τοπικέ κυβερνήσει για να συμφωνήσουμε τι θα να αναπτύσσουμε τα προγράμματα και όταν ε, αυτά έχουν οριμάσει επαρκώ ε, και έχουν επιδεχθεί στο βαθμό που είναι δυνατό οι έξυπνοι στόχοι, τα υποβάλλουμε στι επιχειρησιακέ επιτροπέ για έγκριση. Δεν καθόμαστε στα γραφεία μα εξετάζοντα προτάσει που έρχονται από δεξιά και αριστερά ε, άρα αποφασίζοντας να χρηματοδοτήσουμε ορισμένε και όχι άλλες. Δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση έχουμε δεχθεί αυτό που λέει το ελεκτικό συνέδριο ότι τα έγγραφα για την υποβολή των προτάσεων στις επιτροπές μας σε μάσα θα πρέπει να είναι σαφέστερα. Δηλαδή το πώ παρέχεται η χρηματοδότηση και πώ υποστηρίζονται οι στόχοι του καταπιστευματικού ταμείου, αυτό θα πρέπει να είναι σαφέστερο Όλα αυτά τα έργα που εγκρίθηκαν μέσα στα τρία χρόνια θεωρούμε ότι αποδεικνύουν πως είχε προσθέμενη αξία αποδεδειγμένα το καταπιστευματικό ταμείο ενίσχυσε τον πολιτικό διάλογο και το διάλογο πολιτικής με τις χώρες εταίρους και πράγματι εφαρμόσε καινοτόμες προσεγγίσεις. Αν κάνετε τον κόπο να πάτε στην ιστοσελίδα του καταπιστευματικού ταμείου θα δείτε αποτελέσματα στις εκθέσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ ό,τι έχουμε κάνει για το EDF. Παρέχουμε βασικές υπηρεσίες για 3,3 εκατομμύρια σχεδόν ε, ανθρώπους βάσει ενός ε, υψηλού επίπεδου συστήματο, κάτι που δεν καταφέρουμε να κάνουμε με το EDF. Αυτά είναι κάποια από τα πλέον εκτήματα και κάποια από τα διδάγματα που αποκομίσαμε για το μέλλον. Τα θετικά σχόλια που έχουμε λάβει από τους ενδιαφερομένους μα ε, στι Βρυξέλλε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέρυσι, αλλά και στο επιτόπου επικυρώνει ότι οι επενδύσεις έφεραν καλά αποτελέσματα με το καταπαστευματικό ταμείο και τα υπόλοιπα εργαλεία συνδυάσαμε μακροπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες προσεγγίσεις και βραχυπρόθεσμες προσεγγίσεις για να καλύψουμε τις ανάγκες των εταίρων μας Θα ήθελα επίσης να επαναλαβώ ότι σημειώνουμε τα όσα επισημαίνει το Κοινοβούλιο και το Ελεκτικό Συνέδριο και το επιβεβαιώνουμε τα περισσότερα χρήματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ευρωπαϊκά χρήματα από τους δίκους μας πόρους. Αυτό που δεν έχει συμπεριληφθεί στο ποσό αυτό είναι ότι υπήρξαν πολλά κράτη-μέλη που συγχρηματοδότησαν εκτός του καταπιστεύματος κάποια έργα όπως και άλλοι χορηγοί επίσης ε, συγχρηματοδότησαν τα έργα μας. Καλύτερος έλεγχος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως υπόθηκε ήδη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει στο Συμβούλιο ως παρατηρητής και ε, δεν το ξεχνάμε, το ίδιο θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Είναι ένα ζήτημα που θα συζητηθεί στο πλαίσιο της διακυβέρνησης ε, της νέας περίοδου. Το ζήτημα τώρα της εστίασης στην ανάπτυξη πράγματι πριν από μερικά χρόνια εκπονήθηκαν εκθέσεις ε, που περιλάμβαναν κάποιους ισχυρισμούς ανυπόστατου ε, σε ορισμένες περιπτώσεις το επισημένο σχετικά με αυτό το θέμα. Εμείς πιστεύουμε και αυτό αποδεικνύεται από τι εκθέσεις ε, στην ΟΣΑΤΑΚ ότι οι περισσότεροι οι χρηματοδοτήσεις ότι τα, οι χρηματοδοτήσει έχουν γίνει σωστά όπως είχαν προβλεφθεί. Αν δείτε τα κονδύλια για την ανάπτυξη ε, από ε, όπου και να δόθηκαν ε, χρήματα σε οποιοδήποτε κλάδο είχαν σχέση και με την, αναπτυξιακή, με την αναπτυξιακή προσέγγιση. Φυσικά δεν ζούμε σε ένα τέλειο κόσμο, αλλά προσπαθούμε να βελτιώνουμε τα πράγματα όπου μπορούμε. Ευχαριστούμε. Η DGNIR θέλει να πει κάτι. Η κυρία Γιάκοψεν έχει το λόγο. Thank you, Chair. Thank you, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Κάποιες από αυτές ε, φαίνεται να σχετίζονται στο λόγο της σύστασης του καταπιστευματικού ταμείου σε σχέση με άλλα μέσα. Έχουμε τέσσερα καταπιστευματικά ταμεία, έχουμε ελέγξει τα τρία εξ αυτών και έχουμε αρχίσει να συλλέγουμε κάποια εμπειρία από τα αποτελέσματα του ελέγχου και της λειτουργίας τους. Υπό τη δική μας οπτική, τα βασικά μηνύματα όταν συστήνει κανείς καταπίστευμα δεν είναι να επικαλύψει άλλα μέσα ή διευκολύνσεις, αλλά να δημιουργήσει ένα σύστημα στοχευμένο και συγκεκριμένο ώστε να κατευθυνθεί σε συγκεκριμένους επίσης στόχους. Όπως είχαμε μάθει στο, Μπεκού, στο καταπίθεμα του Μπακού, ήταν, προσπαθήσαμε να αποφύγουμε παράλληλα συστήματα χρηματοδότησης, να αποφύγουμε τις επικαλύψεις, αλλά στοχεύοντας ακριβώς στα συγκεκριμένα έργα. Νομίζω ότι στο καταπίστευμα της Αφρικής σε σχέση με παρουσιακά μέσα βλέπουμε ότι ήταν ε, ταχύτερο, επιτάχυνε τις συμβάσεις, είχε πιο γρήγορες καταβολές σε σχέση με άλλα μέσα και ίσως θα ήταν ενδιαφέρον πώς μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που μπορούν ακόμα και έτσι να επιβραδύνουν την υλοποίηση η οποία πράγματι έχει καθυστερήσει. Δηλαδή η καλύτερη υλοποίηση των έργων. Ως προς τη μεταφορά των κονδυλίων από το EETF είναι πολιτική απόφαση αλλά όταν πράττει κανείς κάτι τέτοιο πρέπει να εξασφαλίζει ότι κινείται προς τις κατάλληλες κατευθύνσεις, σωστούς στόχους και να αποφεύγει τις επικαλύψεις, όπως έλεγα, με άλλα μέσα χρηματοδότησης. Κατά πόσον το καταπίστευμα χρησιμοποιήθηκε για αναπτυξιακούς λόγους, το παράδειγμα βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά έργα που χρηματοδοτούνται. Πρόκειται για ένα μείγμα και αυτό είναι και το αντικείμενο της έκθεσης. Όταν έχει κανείς τόσο ποικίλα έργα, πώς μπορεί κανείς να εστιάζεται στις συγκεκριμένες δράσεις που επιθυμεί και πώς μετρούμε τον αντίκτυπο από τα μεγέθη της Frontex βλέπει κανείς ότι ο αριθμός των ε, παράμων μεταναστών ε, περιορίστηκε, έπεσε, αλλά δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι ο λόγος της μειώση αυτής ήταν το καταπιστευματικό ταμείο και επομένω, αν θέλουμε να επιτύχουμε κάτι πρέπει να είμαστε εστιασμένοι στις προβολές επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας, επιλογής για την συμμετοχή των τοπικών μικαπαόμικρων πρέπει να αντιληφθεί κανείς ότι μιλούμε για ένα δύσκολο πεδίο στο οποίο λειτουργούν και, καθό, και παρότι μάλλον θέλουμε τη συνεργασία τοπικών φορέων υπό την έννοια της ασφάλειας δεν είναι πάντοτε δυνατόν αλλά αυτό που μπορούμε να δούμε από τα δικά μας έργα, από τα έργα που κοιτάξαμε είναι ότι οι τοπικές ΜΚΟ ενέχονται, συμμετέχουν στην υλοποίηση. Και εδώ λοιπόν η στόχευση των τοπικών κοινοτήτων νομίζω ότι εμπίπτει, καλύπτεται. Ε, σας ευχαριστώ η κυρία εισηγήτρια για το κλείσιμο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την κυρία Γιάκοψεν για την τοποθέτησή της. Ε, νομίζω ότι υπάρχουν στοιχεία στα οποία πρέπει να εμβαθύνουμε λίγο παρετέρω. Για την γάμα δελτα ε, συμφωνώ, δηλαδή δέχομαι ότι ε, και εκείνοι δέχονται τις συστάσεις, αλλά παρότι αυτά ανταποκρίνονται σε κάποιες ενθερμό ίσως αντιμετωπίσεις προβλημάτων που είχαμε να αντιμετωπίσει και στο παρελθόν. Η γάμαδελτα ΝΙΑΡ δεν στάθηκε σε θέση να προβλέψει, να κατανοήσει τι ερχόταν και εφόσον δεν φτάσουν σε συγκεκριμένες χώρες αυτό δεν εγγράφεται ως ε, επίγουσα ανάγκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά αυτό δεν με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη. Τώρα τα χρήματα που φαίνεται να λείπουν που είναι και ένα από τα σημεία εστίασης του ελεκτικού συνεδρίου ε, σε αυτό τι γίνεται ε, θα καταβληθούν αυτά που, είχαμε, που είχαν συμφωνηθεί ή όχι και το οποίο σχετίζεται και με τη συγχρηματοδότηση, αλλά μπορούμε να το δούμε και διμερώς με την Κομισιόν ε, και σχετίζονται συνολικά με τη σύσταση του καταπιστεύματος. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνεται εδώ το σημείο αυτό τη ημερησία διάταξη. Καλή σα επιστροφή στο Λουξεμβούργο, κύριε Γιάκοψεν. Και πάμε στο 12 η τόσο πολυπόθητη έκθεση για τη διάθεση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω ΜΚΟ Καλωσορίζω την κυρία Τέρτελμπομ και τις δυνάμεις στο λόγο για να μας τα παρουσιάσει. And, um, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν ξέρω κατά πόσο θα καταφέρετε να δείτε τις διαφάνειες γιατί θα ήταν ε, πιο εύκολο για τους ευρωβουλευτές να με παρακολουθήσουν ενδεχομένω. Να σας πω ποιος είναι ο τίτλος της ειδική μας έκθεση. Διαφάνεια της διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων που εκτελούν οι μη κυβερνητικέ ε, οργανώσεις. Ε, Πετούνται περισσότερες προσπάθειες για την ενίσχυση της διαφάνειας. Θα επικεντρωθώ σε πέντε ερωτήσεις. Γιατί κάναμε αυτό το έλεγχο, τι ερωτήματα θέσαμε, τι μελετήσαμε, τι συστήνουμε και ε, μια σύνοψη στο τέλος των ευρημάτων. Γιατί κάναμε αυτή, αυτό τον έλεγχο. Βασικά αυξάνεται το ενδιαφέρον για τη διαφάνεια στη χρηματοδότηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τις ΜΚΟ για να σχεδιάζει, να εφαρμόζει και να ελέγχει προγράμματα σε πολλούς τομείς πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτελεί γύρω στο 1,7% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και 6,8% του, ε, των ε, Ταμείων Ανάπτυξης μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων. Στη συνέχεια θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες λεπτομέρειες. Και φυσικά υπήρξε κάποια στιγμή και ένα αίτημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γίνει ένας τέτοιος έλεγχος από πλευράς ελεγκτικού συνεδρίου και αν χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια. Για ποιο λόγο λοιπόν διεξήγαμε αυτό τον έλεγχο. Αν δείτε τα αριθμητικά στοιχεία, τι διαπιστώνουμε. Από το 2014 μέχρι το 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμεύσει γύρω στα 11,3 δις ευρώ προς ΜΚΟ. Τα περισσότερα κονδύλια από αυτά αφορούν εξωτερικές δράσεις και κυρίως τομείς όπως είναι η ανάπτυξη που απορροφά το 24%, ανθρωπιστική βοήθεια 26% και στη γειτονία 7%. Βεβαίως, έχουμε και επιδότηση ΜΚΟ για την έρευνα 19%, παιδεία και πολιτισμός 8% και τα υπόλοιπα λοιπά ε, 16%. Στο Λίβανο κάναμε τον έλεγχο ε, στην ανθρωπιστική βοήθεια για τους σύρους πρόσφυγες με ενίσχυση ε, μετρητά. Το έργο αυτό κάλυπτε περίπου 31 εκατομμύρια και επίσης παροχή βοήθεια σε παιδιά και σχολεία για να έχουν περισσότερες ευκαιρίες στην παιδεία και στην υγεία στο Λίβανο, 38 εκατομμύρια περίπου. Για ποιο λόγο λοιπόν κάναμε αυτό τον έλεγχο. Σε αυτή τη διαφάνεια που σας δείχνω εδώ θα σας μιλήσω για τον ορισμό των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Γιατί συνήθως χρησιμοποιούμε τον όρο ΜΚΟ, αλλά δεν υπάρχει ευρέως αποδεκτός και γενικός αποδεκτός ορισμός ε, στις ανακοινώσεις και στις δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ταξινόμηση των ΜΚΟ το 1997. Γίνεται κάποια αναφορά, αλλά υπάρχει και ορισμός που χρησιμοποιούν τα Ηνωμένα Έθνη. γιατί ε, έχουμε εργολαβίες όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από τον ΟΗΕ και δεν είναι ακριβώς η ίδια ε, στην κλιματική κλιμακωτή επιχορήγηση. Συγγνώμη. Τι ρωτήσαμε λοιπόν κατά τον έλεγχο αυτό. Ρωτήσαμε υπάρχει διαφάνεια στη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων από μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Και έχουμε και άλλες υποερωτήσεις. Είναι αξιόπιστη η ε, ταυτοποίηση, μάλλον ο χαρακτηρισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για μία ΜΚΟ. Επίσης, η επιλογή τους είναι κάτι που γίνεται με τρόπο διαφανή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συλλέγει και δημοσιεύει πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτεί τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Τι μελετήσαμε. Αυτό είναι το πεδίο εφαρμογής του ελέγχου το επειδή που ο έλεγχος. Ε, κοιτάξαμε τους κυριότερους τομείς πολιτικής ε, ανάλογα με τον όγκο χρηματοδότησης και τα κονδύλια. Ε, επικεντρωθήκαμε στην εξωτερική δράση. Από το 2014 ελέγξαμε 14 έργα υπό την γίδα των ΜΚΟ, στην άμεση διαχείριση και στην μεικτή διαχείριση την έμεση δηλαδή, έξι έργα. Εξού και ε, έχει τόση σημασία η προηγούμενη διαφάνεια για τον ορισμό. Ε, θα διατρέξω σύντομα τις δύο επόμενες διαφάνειες. Βλέπετε τα κονδύλια που έχουν δοθεί σε ΜΚΟ από το 2014 μέχρι το 2017. Είναι ανάληψη υποχρεώσεων, ε, τα κονδύλια που έχουν δεσμευτεί εκεί, και αν βγάλετε το Ευρωπαϊκό Ταμείο ανάπτυξη, αυτό αντιπροσωπεύει ένα 1,7%. Ε, στην άλλη διαφάνεια ε, βλέπουμε την κατανομή αναγενική διεύθυνση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάλι μπορείτε να διαπιστώσετε ότι αφορά κυρίως την εξωτερική δράση. Τι μελετήσαμε λοιπόν, ποιος ήταν ο στόχος και η προσέγγιση του ελέγχου. Να δούμε κατά πόσο εξασφαλίζεται η διαφάνεια στις συμβάσεις μας ε, με ΜΚΙΟ, γιατί υπάρχει και ευρύτερη διαφάνεια με ποιο τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εντοπίζει και επιλέγει κάποιες ΜΚΙΟ. Γίνεται αυτό με τρόπο διαφανή. Ε, και για την κλιμακωτή επιχορήγηση ισχύει αυτό. Και επίση, όταν έχει κάποια στοιχεία για τις ΜΚΟ τα, τα διασταυρώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα δημοσιεύει με το σωστό τρόπο. Εμείς ε, είχαμε και πολλές συναντήσεις και συνεντεύξεις με ε, υπαλλήλου Ευρωπαϊκή Επιτροπής αλλά δεν κάναμε τον λογιστικό έλεγχο στις ίδιες τις ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Το αφήσαμε αυτό στα χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν ήταν διαφανής ορισμός και η συνεργασία. Και έρχομαι τώρα τα βασικά συμπεράσματα στις παρατηρήσεις αλλά και τις συστάσεις της έκθεσής μας. Πρώτον, Δεν είναι αξιόπιστος ο τρόπος με τον οποίο χαρακτηρίζει κοιό μια οργάνωση ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν εξαρτάται στις περισσότερες περιπτώσεις από το καθεστώς και τη μορφή ε, του νομικού προσώπου. Με τον ίδιο τρόπο ζητούν, ε, κάνουν τις αιτήσει για χρηματοδότηση. και στο λογιστικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν υπάρχει ένα κοινό σύστημα καταχώρησης ε, ε, ετούντων και δεν είναι επαρκή τα κριτήρια ε, με βάση τα οποία χαρακτηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια οργάνωση ΜΚΟ. Είσαι ό,τι δηλώσεις, αρκεί να το δηλώσει η ίδια η οργάνωση, δεν το ελέγχει μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα δεν είναι επαρκώς αξιόπιστη, για να μην πω αναξιόπιστη η διαδικασία αυτή. Κοιτάξτε πώς ταξινομεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια οργάνωση ως μη κυβερνητική. Αρκεί να το δηλώσει η ίδια οργάνωση. Εκείνοι εισάγουν τις πληροφορίες στο σύστημα. Και εδώ βλέπετε τρία διαφορετικά συστήματα, Πάντορ, URF και e-Proposal, υπάρχουν και άλλα. και αυτή τη στιγμή εγκριθεί και χαρακτηριστεί ΜΚΟ μπαίνει στο λογιστικό σύστημα σε ε, επίπεδο ABAC. Στις περισσότερες περιπτώσεις ε, κοιτάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν είναι ιδιωτικές οι οργανώσεις αυτές και μη κερδοσκοπικές και μετά τις καταχωρίζει στο ΑΠΑΚ. Αλλά καμιά φορά μπορεί να είναι πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, ιδρύματα, συνεταιρισμοί κτλ. Τα οποία επίσης χαρακτηρίζουν μη κυβερνητικέ οργανώσεις στο ΑΠΑΚ. Ερχόμαστε τώρα στις συστάσεις. Θα πρέπει να βελτιωθεί ή θα θέλαμε να βελτιωθεί η αξιοπιστία ή το συστήνουμε αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ε, ως προς την ενημέρωση για τις ΜΚΟ θα πρέπει να είναι πιο σαφή, να ορίσουν σαφή κριτήρια μάλλον για το τι είναι μη κυβερνητική οργάνωση και πώς εγγράφεται στο λογιστικό σύστημα, πώς ταξινομείται. Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και αξιοπιστία των μη κυβερνητικών οργανώσεων ως προς την πληροφόρηση που διαδίδεται. Δεύτερη παρατήρηση που οδήγησε στην σύσταση παριθμών 2. επιλογή που γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επίτροπη. Έχουν ε, κάποιες διαδικασίες που μελετήσαμε και είναι γενικά διαφανής, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, διασταυρώνει πολλές φορές τις δηλώσεις για την πρώτερη εμπειρία. Γιατί δεν τα χωράνε ε, τα συστήματα, τα ηλεκτρονικά, όλες αυτές τις πληροφορίες για τη χρηματοδότηση που έχουν λάβουν οι οργανώσεις και τις δραστηριότητε που εκτελούν. Και επίση υπάρχουν διαφορέ ανάμεσα στι διάφορε γενικέ διευθύνσει. Σε τρει περιπτώσει, υπάρχουν οργανισμοί του ΟΗΕ που έχουν χρηματοδοτήσει τρει μη κυβερνητικέ οργανώσει χωρί να ακολουθούν τι ίδιε τι δικέ του διαδικασίε. Ερχόμαστε τώρα στη σύσταση παριθμών 2. Θα πρέπει να ελέγξουν τους κανόνες που ισχύουν και αν ισχύουν για τις κλιμακωτές επιχορηγήσεις, granting. Ε, να ορίσουν κριτήρια για ε, τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτούν τρίτες ΜΚΟ και θα πρέπει να ελέγχουμε κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τηρεί τους κανόνες και τις διαδικασίες. Έρχομαι τώρα στην παρατήρηση παριθμών 3. Οι πληροφορίες που συλλέγονται και δημοσιοποιούνται σχετικά με την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση σε ΜΚΟ. Ο τρόπος με τον οποίο συλλέγονται αυτές οι πληροφορίες δεν είναι ομοιόμορφος. Και στην εξωτερική δράση υπάρχουν περιπτώσεις με ελλειπή πληροφόρηση έως και ε, λανθασμένη. Ε, κυρίως αυτό αφορά η διεθνής ΜΚΟ και ε, έργα όπου, όπου έχουμε έμεση διαχείριση. Τι γίνεται με τη δημοσιοποίηση και την αποκάλυψη των στοιχείων Όλα αυτά γίνονται μέσω του συστήματος ε, οικονομικής διαφάνειας, όπως λέει ο αντίστοιχος κανονισμός, αλλά και πάλι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις διάφορες γενικές διευθύνσεις και όλο αυτό δεν γίνεται πιο διαφανές τελικά. Ε, αυτό μας οδήγησε στη σύσταση παριθμών 3, όπου συστήνουμε να βελτιωθεί η ενημέρωση για τα κονδύλια που διαχειρίζονται ΜΚΟ και έχουμε δύο υποσυστάσεις να βελτιωθεί το σύστημα χρηματοδότησης όλων των δικαιούχων, όχι μόνο των βασικών ΜΚΟ, και επίσης θα πρέπει να βελτιώνεται η χνηλασιμότητα στην εξωτερική δράση, ιδιαίτερα όταν συμμετέχουν διεθνείς ΜΚΟ και φορείς των Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχει και η σύσταση παριθμών 4, η τελευταία κυρία Πρόεδρε, που λέγει ότι χρειάζεται τυποποίηση και βελτίωση ε, της ακρίβειας των πληροφοριών που δημοσιεύονται. Θα πρέπει να αποκαλύπτονται τα ονόματα των δικαιούχων οργανώσεων με το ναι. αντίστοιχο ποσό κάθε φορά. Γι' αυτό αφορά και ιδιαίτερα την εξωτερική δράση. Θα πρέπει να εξακριβώνουμε κατά πόσο οι οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών, ε, διάφορες υπηρεσίες ανταποκρίνονται στο ρόλο τους. Βασικό μας μέλημα είναι η διαφάνεια. Το κοινό δεν ενημερώνεται με τρόπο ουσιαστικό, ε, ούτε γίνεται αναφορά και έκθεση, ούτε καν ε, αναφέρονται τα κονδύλια που έχουν λάβει, με ποιο τρόπο τα έχουν διαχειριστεί, ε, τι γίνεται με τα δίκτυα των διεθνών ΜΚΟ. Συνοψίζω τα ευρήματά μας καταλήγουν σε τέσσερις βασικές συστάσεις, αυτές που σας ανέφερα. Θέλω να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί ήταν πάρα πολύ καλή η συνεργασία μας. εδέχθηκαν όλες τις συστάσεις μας, εκτός από την πρώτη. Πάντως νομίζω ότι είχαμε πάρα πολύ αγαστή συνεργασία και ελπίζω η έκθεση αυτή να βοηθήσει ε, για να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτούνται οι ΜΚΟ και διαχειρίζονται τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μέσω του συστήματος ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επαναλαμβάνω, έγιναν όλα αυτά. Εμεί δεν κάναμε λογιστικό έλεγχο στις ίδιε ΜΚΟ. Πραγματικά, ξέρετε πόσο καιρό δουλεύουμε σε αυτά τα θέματα και πόσο καιρό περιμένουμε. Ε, και εμείς δεν έχουμε τίποτα με τις ΜΚΟ, αλλά θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια και να ισχύει για όλους. Η συγκήτριά μας είναι η κυρία Κλάοντια Σμιτ. Παρακαλώ, ευχαριστώ πολύ. Υποστηρίζω προφανώς όλα αυτά που λέτε. Και τώρα να γίνω λίγο κακιά. Μας έφερε αυτή την ειδική έκθεση το ελεγκτικό συνέδριο και είχα μπει στον πειρασμό να πω ότι το καλό πράγμα αργεί να γίνει, γιατί περιμέναμε πάρα πολύ μέχρι να φτάσει η έκθεση. Αλλά ποιο είναι το καλό πράγμα που αργεί να γίνει, αν δούμε τι έχει διαπιστώσει η ε, ε, ε, έκθεση του Συμβουλίου, του συνεδρίου μάλλον. Μας παρουσίασε την έκθεση τώρα η κυρία Τόρτελμπομ, την ευχαριστώ. Κατά την άποψή μου η έκθεση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει κάτι που φοβόμασταν από καιρό και τώρα, το βλέπουμε γραμμένο στο χαρτί. Τα γεγονότα είναι αμήλικτα και σαφέστατα. Και δεν βοηθάει το να επενείτε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέλος για την καλή συνεργασία. Ε, το πιο ενδιαφέρον ήταν να ακούσουμε ε, με πόση επιπολαιότητα, αν και νόμιμα, διαχειρίζονται κάποια ευρωπαϊκά κονδύλια. Μας λένε ότι τα κριτήρια είναι αρκετά αδιαφανή για να μην βγουν ε, κάποιες μη κυβερνητικές ε, οργανώσεις από τον κατάλογο. Μα αυτοί που τα γράφουν αυτά έχουν χειριστεί κανένα τέτοιο σύστημα διαφάνειας. Για τα κριτήρια επιλογής υπάρχει η κατηγορία ΜΚΟ. Αν κάποιος θέλει και έχει αρκετή υπομονή, μπορεί να κοιτάξει τις ομάδες των δικαιούχων αυτές. Και θέλω να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτές οι κατηγορίες ισχύουν ε, μόνο όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αποδείξει πόσο κοντά είναι στους Ευρωπαίους πολίτες ή και όταν θέλετε να ελέγξετε πολύ προσεκτικά της ΜΚΟ. Αν επιμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το επιχείρημα ότι δεν αρκεί κάποιος να λέει ότι είναι ΜΚΟ για να παίρνει κοινοτικά χρήματα. Ωραία, πώς εξασφαλίζεται ότι ε, είναι όλα σύνομα, ε, τύπικά και λογοδοτούν. Ε, μην μας πείτε ότι δεν υπάρχει νομική βάση στο δημοσιονομικό κανονισμό ε, για να φωτίζει ε, ιδιαίτερα τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Ας πούμε η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που είναι ο υψηλότερος στόχος και αυτό θα πρέπει να γίνεται και η πραγματικότητα. Γιατί αυτό το λένε και οι συνθήκες και το κατοχυρώνουν για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σύστημα μεταφοράς κεφαλαίων, αυτό το FTS, ε, δεν λειτουργεί σωστά μέχρι να μάθουμε ποιος είναι ο τελικός δικαιούχος και πώς ε, ε, χρησιμοποιεί τα κονδύλια αυτά. Τι θα κάνουμε τώρα, θα φεθούμε στην καλή βούληση και ε, στον πατριωτισμό των ε, οργανώσεων αυτών. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχει περιορισμένα και μόνο τα όσα οι ίδιοι δηλώνουν. Καλό είναι βεβαίως επιτόπου να χρηματοδοτούμε τους δικαιούχους και τους εταίρους μας, οι οποίοι ξέρουν τι χρειάζεται η αναπτυξιακή βοήθεια και η ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό που δεν έχει όμως κανένα νόημα είναι να μην παρακολουθούμε πού πηγαίνουν τα κονδύλια αυτά. Και αυτά που ακούω για τα απόρριτα, τα εμπιστευτικά και τα ζητήματα ασφαλείας, τα ακούω βέρεσε. Λοιπόν, αρκετά ε, σας τα έψαλα και με κοιτάτε όλοι ε, έτσι περίεργα. Το θέμα είναι πού είναι τα ευρωπαϊκά κονδύλια και πώς ελέγχονται, γιατί πρέπει να ελέγχονται. Και έχει έρθει η ώρα να ανταποκριθεί στο ρόλο της ε, ως θεματοφύλακας των συνδικών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριος Νίντα Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα κάνω δύο σύντομα σχόλια, αλλά πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω το ελεκτικό συνέδριο για τις προσπάθειες του, το έργο του, για τις τέσσερις συστάσεις και την εκθέση αυτή. Γνωρίζω ότι η Επιτροπή μας ζήτησε την ειδική έκθεση για την διαφάνεια των ευρωπαϊκών κονδυλίων που παρέχονται στη ΜΚΟ. Η ερώτηση που θέλω να κάνω είναι η εξής. Αν αυτή η προσέγγιση μεθοδολογικά είναι σωστή και αν σχεδόν όλα τα ευρήματα σε αυτή την ειδική έκθεση θα πρέπει ε, ενδέχεται να μην ισχύουν για όλους τους άλλους δικαιούχους ε, πέραν των ΜΚΟ. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι υπάρχει λόγος να εστιαζόμαστε μόνο στις ΜΚΟ όσον αφορά τη διαφάνεια των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Το δεύτερο που θα ήθελα να σχολιάσω εδώ εν συντομία, όταν αξιολογούμε τους ετούντες και τα έργα θα πρέπει να εστιαζόμαστε στο πώ συνάδουν τα έργα με του προγραμματιζόμενου στόχου και πώ οι στόχοι έχουν επιτευχθεί εντό των έργων. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε περισσότερο διοικητικό φόρτο στι ΜΚΟ από αυτό που μπορούν να αντέξουν. Αυτό ισχύει ειδικότερα για τι ε, ΜΚΟ που άμεση αντίδραση σε ανθρωπιστικά θέματα. Η αναθεώρηση του χρηματοοικονομικού κανονισμού απλούστευσε του κανονισμού, του κανόνες, συγγνώμη. Αυτό έγινε ευπρόσδεκτο από όλου του δικαιούχου. Δεν πρέπει να οπισθοδρομήσουμε. Σήμερα οι ΜΚΟ αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις παγκοσμίω. Δυστυχώ και σε ορισμένα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι ΜΚΟ στη διατήρηση της συνοχής της κοινωνίας σε σημαντικούς τομείς πολιτικής όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η παιδεία, τα περιβαλλοντικά ζητήματα και οι κοινωνικές πολιτικές. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να πω ότι ναι, η διαφάνεια μεν είναι πάντα ευπρόσδεκτη, αλλά εντός λογικών ορίων. Η ελευθερία δράσης των ΜΚΟ είναι επίσης ύψης της σημασίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Στάς, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, άκουσα τον κύριο Νίτερ Μιουλέρ. Θέλω να καλωσορίσω εδώ την κυρία Τέρτερμπορ. Ε, είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην Επιτροπή μας και η πρώτη ειδική έκθεση που μας παρουσιάζει. Καλωσορίσατε και χαίρομαι που ήρθατε. Συνεχίζω από εκεί που σταμάτησε ο κύριος Νίτερ Μιουλέρ. Έχει μεγάλη σημασία η διαφάνεια, χωρίς καμιά αμφιβολία και θα πρέπει να φροντίζουμε όλα να γίνονται με σωστό τρόπο αλλά να μην οδηγούν όλα αυτά ε, στο να ζητάμε τον ουρανό μετάστρα ε, και να έχουμε υπερβολικές απαιτήσει από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Ένα αυτό. Δεύτερον, φαίνεται από τη συζήτηση, πώς να το πω, λες και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις παίρνουν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν ελέγχονται καθόλου ή δεν ελέγχονται παρκώ για το πώ τα δαπανών. Άκουσα στην εισαγωγή τη την κυρία Τέρτολμπαμ να λέει ότι αυτή η ειδική έκθεση δεν μιλάει για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων από τις ΜΚΟ, τα συστήματα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξασφαλίζει τη διαφάνεια. Αυτό είναι το αντικείμενο. Και σας ερωτώ, μετά από τη δουλειά που κάνατε εσείς με τους συνεργάτες σας, μπορείτε να πείτε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει έλεγχος ή υπάρχει ανεπαρκής έλεγχος ε, στα κονδύλια που διαχειρίζονται ΜΚΟ για να ε, υλοποιούν κάποιους από τους στόχους. Αυτό μπορούμε να το συνάγουμε από την δική σας ειδική έκθεση, γιατί αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε δεν χρειάζεται να ε, υποδιόμαστε εδώ και να συνεχίζουμε να υποδιόμαστε ότι δεν υπάρχει έλεγχος, γιατί έρχεται να το αποδείξει η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Έχω γράψει και εγώ το όνομά μου στον κατάλογο των ομιλητών, λέει η Πρόεδρος. Και θα σας παρακαλούσα ε, να καταλάβουμε ότι η συζήτηση εδώ δεν είναι αν είμαστε υπέρ ή κατά των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Και δεν θέλω τώρα να στριμώξω κανέναν σε ένα κράτος μέλος, που είναι έτσι κι αλλιώς δύσκολη η κατάσταση, να μην την επιβαρύνουμε περισσότερο. Αυτό όμως που θα πρέπει να αναρωτηθούμε είναι πόσα χρήματα πηγαίνουν σε ΜΚΟ και ακούσαμε από τη μελέτη και την επόμενη που θα ακούσουμε είναι επίσης πολύ ενδιαφέρουσα γιατί είναι μαύρο κουτί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν διοίκηση δική της. Τα κράτη-μέλη έχουν κρατικές διοικήσεις και χρειάζονται ε, και συμπλήρωση και βοήθεια και όπου δεν έχουν αυτή τη βοήθεια την αναθέτουν σε εξωτερικούς και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς φτάνουμε στους στόχους πολιτικής για την εκτέλεση των πολιτικών μας δια των ΜΚΟ. Αυτό δεν το ψάξατε, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι ΜΚΟ τι σκοπούς εξυπηρετούν και πολιτικούς δικούς τους, ίδιους ε, ε, ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το ερώτημα κρύβεται από πίσω και προσπαθήσαμε επανειλημμένα εδώ στην Επιτροπή μας με πολλές μελέτες να κατανοήσουμε, να συλλάβουμε. Αλλά εμένα με εκπλήξει κάθε φορά που ρωτάμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά από λίγα χρόνια κάτι άλλο, βγαίνουν τελείως διαφορετικά αριθμητικά στοιχεία. Και τώρα θα πρέπει να ορίσουμε κάποια στιγμή τι εστί ΜΚΟ. Και αν δεν το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα το κάνω εγώ το αργότερο στην αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού. Ε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να μην... Ε, ε, έχουμε ένα εισοδισμό πούμε, και να μπαίνουν στην κατηγορία μήκη όργανος που δεν έχουν καμιά δουλειά να βρίσκονται εκεί. Εμείς κάναμε πάρα πολλά για ΜΚΟ, απεμπολίσαμε την προοδευτική μείωση, ε, τη σταθερότητα, διάφορα κριτήρια και καταλαβαίνουμε ΜΚΟ ότι τις εκτιμούμε. Αλλά το τι κάνουν πρέπει να το ελέγχουμε και στην εμπορική πολιτική μπορεί ο καθένας να έχει άλλη άποψη. Αλλά τώρα εδώ πρέπει να χρηματοδοτούμε ε, μη κυβερνητικέ οργανώσει που είναι κατά του ελεύθερου εμπορίου. Μα τι έγινε, μα έχει στρίψει τελείω. Ε, ο στόχο μα είναι η εμπορική πολιτική, όχι η παρεμπόδιση τη εμπορική Γιατί έτσι ξεκινάνε σιγά σιγά διάφορε καταστάσει και περιεργίες. Και πρέπει να σα πω ότι δεν σταματάει σήμερα εδώ. Έχουμε όμω και άλλο θέμα στη μέση διάταξη, γι' αυτό θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α, δεν ξέρω. Είναι και άλλη συνάδελφοι. Α, είναι. Σαγιάλα ήθελε εκεί το λόγο. Ναι, πρόεδρε. Καταρχάς, να καλωσορίσουμε το Ευρωπαϊκό, το Ελεκτικό Συνεδριό που έχει κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά υπό τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Γνωρίζουμε τα θέματα αυτό ότι δεν είναι ουδέτερα και εύκολα τα σχετικά με την ΜΚΟ, της ΜΚΟ, αλλά έχουμε λάβει κατάλογο επιχειρήσεων που βρίσκονται και εισηγμένες και τις οποίες χρηματοδοτούμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι ΜΚΟ έχουν ε, μια πολύ πιο άμεση επαφή με τους πολίτες από επιχειρήσεις άλλες. Ευχαριστώ λοιπόν την κυρία Τρότελμπούμ για τη δουλειά της, αλλά εδώ προσπαθούμε να εξετάσουμε υπό ποιο σύστημα οι μη έχουν πρόσβαση σε κονδύλια υπό τις εντολές και τους στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της μετανάστευσης, ε, στο πλαίσιο των προσφύγων και χάρη στις οποίες ε, τελικώς καταφέρνουμε να φτάσουμε Στου τελικού δικαιούχου που θέλουμε να ενισχύσουμε. Τώρα, είναι προφανές ότι οι οντότητε ε, που δουλεύουν για άλλα συμφέροντα, για να προασπίσουν άλλα συμφέροντα, δεν θα έπρεπε καθόλου να βρίσκονται στον κατάλογο των καπαόμικρων και πολύ περισσότερο στον κατάλογο των καπαόμικρων που ενισχύουμε εμείς. Και η κυρία Τρόιτλμπούμ... Ε, εδώ υποβάλλει μια πρόταση με μεγέθη και δεδομένα Υπάρχει τα θέματα του ορίζοντα 2020, τα θέματα ασφαλείας, ε, κοινωνίας των πολιτών, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Είδαμε βέβαια ε, να επανεθνικοποιούνται πολλοί στόχοι και κατευθύνσεις και με ανησυχεί κάπως το γεγονός ότι τελευταία χρόνια είδαμε ότι κάποιες από τις οργανώσεις που πραγματικά είχαν ευρωπαϊκή εμβέλεια και που είχαν λειτουργήσει στα πλαίσια ευρωπαϊκών συγκρούσεων και που ήταν οι μοναδικές που μπορούσαν να υποστηρίξουν και να υλοποιήσουν πραγματικά αυτές τις, δράσεις, τις ευρωπαϊκές δράσεις αντικαταστήθηκαν σταδιακά από οργανώσεις τελικώς εθνικής, εθνικού χαρακτήρα. Ε, κάθε κράτος μέλος έχει μια δική του προτιμητέα μη καπαόμικρον ε, με, για την προάσπιση συμφερόντων που δεν είναι εν πάση πανευρωπαϊκά αναγκαστικά σε κάθε περίπτωση ή σε όλες τις περιπτώσεις. η, αρχική μας στόχευση ήταν η βοήθεια των μη καπαομίκρων που είχαν πραγματικά πανευρωπαϊκή στόχευση, εμβέλεια, λειτουργία. Και δεν έχουμε εδώ ε, καμία δουλειά να ενισχύουμε στόχους που εν πάση εκτός δεν έχουν σχέση με το ευρωπαϊκό όραμα. Εγώ αυτό ήθελα να ακούσω λίγο από την Κομισιόν. Ε, αυτά που μας λέει η κυρία Τρούτλμπούμ είναι, είναι σε ένα προηγούμενο στάδιο και την ευχαριστώ για τη δουλειά αυτή αλλά θα μου αρέσει να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν κατά πόσο αναλυθεύει αυτή η εντύπωση που έχουμε και που είναι αυξανόμενη ότι αυτές οι οργανώσεις που είχαν ένα πανευρωπαϊκό όραμα και εμβέλεια αντικαθιστούνται σιγά σιγά από πιο στενά εθνικές μικρα μικρών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιάλα μου Με παρακάλεσε ο Πρόεδρος να προεδρεύσω εγώ γιατί χρειάστηκε να βγει για λίγο έξω. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Ροζαλτέα Μπρουσκέτς από τη Γενική Διεύθυνση Προπολογισμού. Πού κάθεστε? Hello, Sie haben das Wort. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Uh, thank you, Chair. Hello, everybody. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλους, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο για αυτές τις εκθέσεις Συζητήσαμε πολύ μαζί τους σε ολόκληρη τη διαδικασία του ελέγχου. Έχουμε συμφωνήσει επί πολλών σημείων, αλλά όχι επί όλων. Δεν έχουμε γραφτεί συμφωνία. Σήμερα εδώ υπογραμμίσατε διάφορα ζητήματα. Ξεκινώντας, θα ήθελα να πω ότι ο έλεγχος αυτός αφορά τη διαφάνεια όσον αφορά τις ΜΚΟ. Δεν αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι ΜΚΟ υλοποιούν τα προγράμματα, ούτε αφορά τους ελέγχους ε, που ε, εκτελεί η Κομισιόν σχετικά με αυτό. Πρέπει να πω ότι η Κομισιόν πραγματοποιεί όλου του ελέγχου όπω έχουν προβλεφθεί στο χρηματοοικονομικό κανονισμό, όχι μόνο για τις ΜΚΟ, αλλά και για όλου του οργανισμού και για όλους τους δικαιούχους που υλοποιούν τον ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό λίγο πιο επί της ουσίας των ελέγχων αυτών. Θα σας εξηγήσω τα οριζόντια θέματα και υπάρχουν και συναδελφοί από τις Γενικές Διευθύνσεις ΝΙΑΡ, και ΕΚΟ και αν έχετε πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις μπορούν να τις απαντήσουν. Ήθελα να πω ότι στην έκθεση πολλά ευρήματα βρίσκουν σύμφωνοι την Κομισιόν. Ως απάντηση σε αυτή την έκθεση, στην Κομισιόν έχουμε εξηγήσει ότι γίνονται διαρκείς προσπάθειες διασφάλισης της διαφάνειας. Έχει δεσμευτεί με αυτό η Κομισιόν να διασφαλίζει την διαφάνεια. Πιστεύουμε ότι είμαστε ένας από τους οργανισμούς παγκοσμίω ε, που παρέχει πολλές πληροφορίες για το ποιος και πώς ε, υλοποιεί τον προϋπολογισμό. Το ελεκτικό συνέδριο έκανε τέσσερις συστάσεις και η Κομισιόν δέχθηκε τις τρεις. Να σας διευκρινίσω τι έχει γίνει για την καθεμία. Ξεκινάω με τα σημεία επί των οποίων συμφωνούμε. Η πρώτη σύσταση με την οποία συμφωνούμε είναι οι δύο. Σε αυτήν το ελεγκτικό συνέδριο συνιστά στην Επιτροπή να εφαρμόζει όλους τους ε, κανόνες κλιμακωτής ε, επιχορήγησης λαμβάνοντας υπόψη τις τομεακές ιδιαιτερότητες. Πρέπει να πω ότι δεχόμαστε αυτή τη σύσταση και πράγματι θεωρούμε ότι έχει ήδη αναλυφθεί η δράση με τις αλλαγές που εισήχθησαν στην τελευταία εκδοχή του χρηματοοικονομικού κανονισμού. το χρηματοοικονομικό κανονισμό, στον νέο χρηματοοικονομικό κανονισμό, δημοσιονομικό κανονισμό, έχουμε σαφείς κανόνες που εφαρμόζονται υποχρεωτικά από όλους τους ενδιαφερομένους. Όσον αφορά τη σύσταση 3, Το ελεγκτικό συνέδριο συνιστά στην Επιτροπή να βελτιώνει τις πληροφορίες που λαμβάνει για τα χρήματα που λαμβάνουν με τα διάφορα συστήματα επιχορήγησης ή ΜΚΟ. Έχουμε ήδη βελτιώσει πολύ τα πράγματα στον τομέα της έρευνας. Παλιότερα δημοσιοποιούνταν μόνο οι πληροφορίες για τους συντονιστές στα σχετικά συστήματα. Τώρα στον τομέα της έρευνας παρέχουμε πληροφορίες όχι μόνο για τον συντονιστή, αλλά και για όλους τους συνδικαιούχους των ε, Ταμείων της Ένωσης. Σε όλους τους τομείς ε, πραγματοποιούμε μια ανάλυση για να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα συστήματα διαχείρισης στο μέλλον, ώστε να μπορούμε να συλλέγουμε όλες τις πληροφορίες, ε, ειδικότερα για την εξωτερική δράση και Προσπαθούμε να αλλάξουμε τις συστήματα διαχείρισης που υπάρχουν, ώστε να διαχειρίζονται καλύτερα αυτά τα κονδύλια και να είναι ε, διαθέσιμες σε πληροφορίες που αφορούν όλα τα βήματα υλοποίηση του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τη σύσταση 4, το Ενεκτικό Συνέδριο συνιστά στην Κομισιόν να βελτιώσει την ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιοποιούνται. Η Κομισιόν θα ήθελε να τονίσει ότι έχουμε δεσμευτεί για τη διαφάνεια πλήρως. Έχουμε ξεκινήσει να αναλαμβάνουμε και δράσεις στον τομέα. Πρώτα απ' όλα αρχίσαμε να δημοσιοποιούμε στο πλαίσιο της ε, διεθνούς πρωτοβουλίας ε, για τη διαφάνεια της ε, υποστήριξης στοιχεία για τις βοήθεια που παρέχουμε και το 2015 και το 2017 ε, έχουμε αναλύσει λεπτομερώς ε, φυσικά όλες τις συστάσεις ε, του ελεκτικού Συνειδρίου και θα αναλάβουμε και άλλες δράσεις που θα καταστούν απαραίτητες. Κάτι άλλο για το οποίο επέμεινε το Ελεκτικό συνέδριο αφορά την έμεση διαχείριση. Όταν τα κονδύλια χρησιμοποιούνται από οργανισμούς των ΗΕ για παράδειγμα. Από αυτή την άποψη, καλό θα ήταν να πούμε ότι στο πλαίσιο της έμεσης διαχείρισης το σύστημα της ε, αξιολόγησης εξάντε ε, βοηθά την Κομισιόν να βασίζεται στα εργαλεία και στις διαδικασίες αυτών των έμπιστων οργανισμών. Όλες αυτές οι αξιολογήσεις πυλώνων, όπως ονομάζονται, έχουν εισαχθεί και στο δημοσιονομικό κανονισμό. Αυτέ είναι οι τρει συστάσει που έχει δεχθεί η Κομισιόν. Αλλά όπως είπα, για την πρώτη σύσταση είναι δυνατόν να δεχθούμε την σύσταση του την πρώτη σύσταση συγγνώμη, του δικαστηρίου. Γιατί, Γιατί αυτή η πρώτη σύσταση του, του ελεγκτικού συνεδρίου συγγνώμη, λέει ότι η Κομισιόν θα πρέπει να βελτιώσει το λογιστικό σύστημα με σαφείς εσωτερικές οδηγίες και σαφή κριτήρια ταυτοποίησης των ΜΚΟ και προσδιορισμού των ΜΚΟ. Εδώ θα πρέπει να είμαστε σαφεί. Η Κομισιόν θέλει διαφάνεια, αλλά δεν υπάρχει κοινό ορισμό των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Και δεν μπορεί κάτι τέτοιο να λυθεί με το λογιστικό σύστημα. Εγώ είμαι υπεύθυνη για το λογιστικό σύστημα, είμαι αξιωματούχο λογιστική τη Κομισιόν. Δεν είμαι εγώ αυτή που θα καθορίσω, θα δώσω τον ορισμό τη ΜΚΟ. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει σαφής ορισμό. Υπάρχουν ορισμοί σε κάποια κράτη-μέλη, αν βάλω εγώ στο λογιστικό σύστημα κριτήρια προσδιορισμού των ΜΚΟ, την επόμενη μέρα θα με κατηγορούν που συμπεριέλαβα τέτοια κριτήρια και όχι κάποια άλλα. Πριν από μερικά χρόνια το Κοινοβούλιο, διότι τέθηκε αυτό το ζήτημα του ορισμού των ΜΚΟ, ζήτησε από την Κομισιόν να πει τι είναι ένας μη ε, μια, μια μη κυβερνητική οργάνωση και τι είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση. και εμείς ε, τότε προσαρμόσαμε ανάλογα τα κεντρικά μας συστήματα για να συμπεριληφθούν αυτές οι πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες είναι δύσκολο να επαληθευτούν. Και για όλους τους δικαιούχους ε, που έχουν εγγραφεί στα κεντρικά συστήματα ελέγχουμε αυτές τις πληροφορίες. Αλλά για τις ΜΚΟ, εφού δεν υπάρχει ορισμός μου, είναι αδύνατο να επαληθεύσω αν ε, μια οργάνωση είναι μη κυβερνητική ή όχι. Αλλά επειδή όλοι μιλάνε για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, έχουμε ε, λαμβάνουμε υπόψη τις ε, δηλώσεις των ίδιων των δικαιούχων. Ζητάμε δηλαδή από τους δικαιούχους των ευρωπαϊκών κονδυλίων να μας λένε αν είναι ιδιωτικές εταιρείε με κερδοσκοπικές και μπορούν να κάνουν μια δήλωση με την οποία δηλώνουν ότι είναι μικρό στα δικά τους ε, κράτη, στα οικία κράτη-μέλη. Αυτή την πρωτοβουλία την πήραμε πριν από μερικά χρόνια. Αλλά αυτή η δήλωση από τι οργανώσει αυτέ είναι δυνατόν να επαληθευτεί αφού δεν υπάρχουν κριτήρια. Η Κομισιόν θεωρεί ότι οποιαδήποτε περαιτέρω κριτήρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα απαιτούσαν εναρμόνιση τη έννοια τη μη κυβερνητική οργάνωση που θα πρέπει να συμφωνηθεί από του νομοθέτε και δεν μπορεί να εισαχθεί απλά από την Κομισιόν για να κλείσω, αναγνωρίζουμε τις μη κυβερνητικές οργανώσεις σίγουρα ως ε, σημαντικούς ε, ε, υποστηρικτές ε, της διακυβέρνησης και των προγραμμάτων αρρωγής και θέλουμε να τις υποστηρίζουμε. Επιπλέον η Κομισιόν είναι ένας από τους πιο διαφανείς οργανισμούς στον κόσμο, ανεξάρτητα από το αν το θέμα αφορά τις δικές μας πρακτικές ή το, η συνεργασία μας με άλλους περαιτέρω βελτιώσεις φυσικά είναι πάντα ε, ευπρόσδεκτες και οι συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου θα μας βοηθήσουν από αυτή την άποψη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Αυτό το θέμα με τη διαφάνεια θα το ξαναδούμε τώρα. Η κυρία Τόρτελμπομ και μετά ο συνάδελφος Ντόιτς. Παρακαλώ. Um, uh, first of all, I would... Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να τονίσω ότι ο έλεγχος δεν αφορούσε στα αποτελέσματα των έργων. Και η συνάδελφος η κυρία Γιάκοψεν ήταν υπεύθυνη για πάρα πολλές ειδικέ εκθέσεις όπου πήγαμε στις λεπτομέρειες των έργων, στα παραδοντέα κτλ. Και είναι σημαντικό αυτό. Το είπα στην εισαγωγή μου, ήθελα να το επαναλάβω. Όμως ο δικός μας έλεγχος ήταν σχετικά με το να καταλάβουμε ποιος κάνει τι και τι ενίσχυση λαμβάνει ο καθένας και πώς δημοσιοποιούνται αυτές οι πληροφορίες. Ελέγχοντας λοιπόν τα διάφορα συστήματα είδαμε ότι για παράδειγμα υπάρχει αυτό το σύστημα ε, λογιστικής δεδουλευμένων ABAC όπου καταχωρίζονται οι οργανώσεις ως μη μικρών χωρίς να υπάρχει σαφής ορισμός. Εμείς λοιπόν για αυτό το λόγο βάλαμε τη σύσταση που λέμε τοποθετώντας το άμπακ στη λογιστική άμπακ χωρίς σαφή ορισμό είναι μια έλλειψη. Καλύτερα θα ήταν να έχουμε μια, έναν ορισμό. Γιατί έχουμε και άλλες περιπτώσεις που ονομάζουμε οργανώσεις μη δεν λέμε τώρα ότι εκείνες δεν χρησιμοποιούν σωστά τι πληροφορίε, αλλά θα ήταν πολύ σαφέστερο να γνωρίζουμε τι περιεχόμενο πρέπει να έχει με ένα φορέας ώστε να ονομάζεται μη Θα ήταν προ το συμφέρον όχι μόνο των Ευρωπαίων φορολογουμένων, αλλά και των ίδιων των οργανώσεων που λαμβάνουν χορηγίε, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά από τα κράτη-μέλη, ιδιωτικέ χορηγίε κτλ. Αυτό ήταν ο λόγος που το είπαμε. Τώρα, κάθε αυτή, καθε αυτη καθε αυτή οι μη δεν είναι πιο επικίνδυνοι δικαιούχοι από άλλη ομάδα, από άλλη κατηγορία. Αλλά υπό την οπτική της ΙΕΔ, εδώ διοχετεύουμε κονδύλια σε διάφορα επίπεδα μη κυβερνητικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων φορέων των ΗΕ ή συμπράξεων με ομικρόν. Και εδώ υπάρχει ένα κίνδυνος ελλειπού διαφάνειας. Στην εισαγωγή μου έδωσα το παράδειγμα που είδαμε σε κάποιες περιπτώσεις ελέγχου, περιπτώσεις με οργανώσεων που δεν καλουθούν τους ίδιους τους τους κανόνες ή τους ίδιους τους τους ορισμούς. Και επομένως στην άμεση ενίσχυση μάλλον στην άμεση διαχείριση ή στην έμεση διαχείριση, αυτό διαφοροποιεί τελείω το πράγμα και καλό θα ήταν να ξέρουμε τι από τα δύο είναι. Θα ήταν προ το συμφέρον όλων να έχουμε περισσότερη διαφάνεια. Νομίζω ότι απάντησα έτσι όλες τις ερωτήσεις. Αν έχω ξεχάσει κάτι, παρακαλώ να μου το θυμίσετε για να επανέλθω ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με την Πρόεδρο. Ότι ε, τα θέματα ουσίας δεν είναι του παρόντος και δεν πρέπει σήμερα να τα λύσουμε, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπούμε και σε θέματα ουσίας για το συγκεκριμένο θέμα. Τι γίνεται με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί για τα ποσά δεν είναι ευκαταφρόνητα, είναι δισεκατομμύρια. Και κατά περίπτωση ε, αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τα κράτη-μέλη, αλλά πρόκειται για ε, χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Κάποια στιγμή να τα συζητήσουμε και αυτά έτσι επί της ουσίας. Ας πούμε, τι γίνεται με τις συγκεκριμένες μη κυβερνητικέ οργανώσεις που αντιστρατεύονται το παγκόσμιο εμπόριο και τι τις χρηματοδοτούμε. Αυτό συνάδει με τις αρχές και τις αξίες μας. Δεν θα πρέπει να μας προβληματίσει. Η δραστηριότητα των μη κυβερνητικών οργανώσεων τα τελευταία χρόνια είναι όντως μη κυβερνητική, γιατί καμιά φορά φαίνονται ε, ε, σαν ημικρατικοί ε, φορείς. Όχι τώρα, αλλά να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ το ελεκτικό συνέδριο για την έκθεσή σας. Με την έκθεση αυτή την ειδική μπορεί να αρχίσει μία διαδικασία ή να δρομολογηθεί, εν περιπτώσει, για να δούμε τα θέματα και στην ουσία τους. για να δούμε τι είναι κυβερνητική οργάνωση, τι είναι μη κυβερνητική οργάνωση και τι ιδιωτική εταιρεία από όλους αυτούς που χρηματοδοτούμε. Αυτό θα πρέπει να ισχύει για όλους. Και η διαφάνεια και οι απαιτήσει ανεξαρτήτως νομικής μορφής. Και στον τομέα των επιχειρήσεων, ε, δεν είναι όλες οι επιχειρήσεις ίδιο. Υπάρχουν μεγάλοι πολυεθνικοί όμιλοι και οικογενειακές επιχειρήσεις. Όλοι όμως οφείλουν να τηρούν τα βιβλία τους με τον ίδιο διαφανή και σωστό τρόπο. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Για σήμερα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι ξεκινάει μια νέα διαδικασία και να ξεφύγουμε από αυτή τη ρητορική που λέει ότι όποιος επικρίνει ε, μια ΜΚΟ για ε, αδιαφάνεια ε, έχει άδικο. Θα πρέπει να τελειώνει αυτή η ρητορική και ελπίζω να περάσουμε σε μια νέα εποχή προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η συγγήτρια για να κλείσει. Κλάουντια Σμιτ. Καλώς. Δεν θέλει. Ωραία. Τελειώνει το σημείο αυτό της μέσης διάταξης. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση της έκθεσης και για την